Uh, Καλημέρα σας. Δυστυχώς ο πρόεδρός μας, ο κύριος Τάνζο έχει κολλήσει στην κίνηση. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρει να έρθει λίγο αργότερα. Κάποιες πληροφορίες να σας δώσω, ανακοινώσεις γλωσσικό καθεστώς. Οι ακόλουθες γλώσσες δεν θα μεταφραστούν. Δανέζικα, φιλανδικά, σουηδικά, λετονικά, σλοβενικά, μαλτέζικα, βουλγάρικα, τσέχικα, σλοβακικά και εσθονικά. Σα ζητώ συγγνώμη. Επίσης σας υπενθυμίζω ότι ε, οι γλώσσες των ε, πληρών μελών έχουν την ε, προτεραιότητα. Επίσης μεταδίδεται ζωντανά η συνεδρίαση αυτή από το διαδίκτυο και εφόσον δεν υπάρχουν ε, αντιδράσεις μπορούμε να εγκρίνουμε τη μερίσια διάταξη και πρέπει να εγκρίνουμε και τα πρακτικά της συνεδρίας της 6ης Οκτωβρίου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ένσταση. Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά. Καλώς ορίσατε για μια ακόμη φορά. Θα δώσω τώρα τον ε, λόγο στον κύριο Πάσκου, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αναφερθούμε σε ένα σημείο στη μερίστη διάταξη σήμερα για το οποίο θα μιλήσουμε για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Αφρική η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η Υποεπιτροπή μας έχουν προσκαλέσει τον πρέσβη Ραμπτάνε Λαμαμρά, Επίτροπο της Αφρικανικής Ένωσης για την Ειρήνη και την Ασφάλεια, καθώς επίσης και τον κύριο Νίκολα Βέστκοτ, που είναι ο εκτελεστικός διευθυντής για την Αφρική στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξ ονόματος λοιπόν της Επιτροπής θα ήθελα να σας καλωσορίσω κύριε πρέσβη Λαμαμρά, καθώς επίσης και τον κύριο Βέστκοτ για τη συζήτηση αυτή που θα έχουμε. Προσβλέπουμε στην συζήτηση αυτή, όπως ξέρετε, μία αντιπροσωπή μας και ο κύριος Γκάλερ ήταν μέλος αντιπροσωπής αυτής, αν όχι επικεφαλής της, επισκέφθηκε την Ίσα και είχαμε και συζητήσεις, κυρίως με εσάς κύριε Πρέσβη, όσον αφορά την κατάσταση στην Αφρική. Θυμάμαι ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίασης που είχαμε εκεί είπαμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Αφρική ως ενιαία ήπειρο και ότι οι συνέργειες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Βόρειας ακτής της Αφρικής καθώς επίσης και των υπόλοιπων περιοχών θα πρέπει να ενισχυθούν. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε ποια είναι η δική σας άποψη για το πώς θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση να συνεργαστούν προκειμένου να προωθήσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα ως προϋπόθεση για την ειρήνη και την ασφάλεια. Επίσης, κύριε Πρέσβη, θα ήθελα να σας ζητήσω να αναπτύξετε λίγο περισσότερο το πώς θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της αποστολής Άμισομ, την οποία επισκεφτήκαμε και στο παρελθόν και σαφώς βέβαια ο κύριος ε, Westcott ε, δεν πρόκειται να γλιτώσει και αυτός από τα αιτήματά μας, γιατί θα χρειαστεί να μας ε, πει ποια είναι η άποψή του για το πώς θα καταφέρουμε να ενισχύσουμε την γενικότερη σχέση που υπάρχει μεταξύ της Αφρικανικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πολύ σημαντική αυτή περιοχή του πλανήτη. Σας ευχαριστώ πολύ και κύριε Πρόεδρε καλωσορίσατε κι εσείς και σας επιστρέφω την Προεδρία. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση αυτή. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Πασκού για τα εισαγωγικά του λόγια. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της, Επιτροπή, της Υποεπιτροπής, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν θα ήθελα εδώ πέρα να ξεχάσω το όνομα κάποιου ευρωβουλευτή, επομένως θα χρησιμοποιήσω την φράση την οποία λέμε και στην Αφρική, στη Δυτική Αφρική, all protocols observed, προκειμένου να απευθυνθώ σε όλους σας. Θα ήθελα λοιπόν να πω κάποια εισαγωγικά λόγια στην αρχή, κάποιες γενικές παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω και θα έχουμε κατά αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα και στη συνέχεια να μιλήσουμε για πιο συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία εσείς θα επιλέξετε για τη σημερινή μας συζήτηση. Καταρχάς όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ θερμά τον κύριο Γκαμπριέλ Μπερτίνη, ο οποίος είναι πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, καθώς επίσης και τον κύριο Αρνό Ντανζό, πρόεδρος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να τους ευχαριστήσω λοιπόν για την πρόσκλησή τους και για τη δυνατότητα που μου δίνουν να συμμετέχω σήμερα σε μια συζήτηση όσον αφορά την εταιρική σχέση και τη σχέση γενικότερα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρικανική Ένωση. Και όλος ιδιαιτέρως θα ήθελα να αφαιρθώ στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Αφρικανική Ένωση στην διαχείριση της ασφάλειας και της ειρήνης στην Αφρικανική Ήπειρο. Θα ήθελα επίσης ε, να ευχαριστήσω και την ε, αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Αντίσα Μπέμπα, η οποία λειτουργεί παράλληλα και συμπληρώνει ουσιαστικά και την αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης ε, στις Βρυξέλλες και κατά αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια πολύ στενή διασύνδεση ανάμεσα στις δύο αυτές οργανώσεις, στα δύο αυτά θεσμικά όργανα, τα οποία φιλοδοξούν να υλοποιήσουν τα πολύ σημαντικά προγράμματα τα οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έχουν αποφασίσει στις συνόδους αυτές, οι οποίες δημιούργησαν τις προποθέσεις για μια βιώσιμη εταιρική σχέση ανάμεσα στην Αφρική και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα επίσης ε, να πω ότι ε, ο διάλογος ανάμεσα στην Αφρικανική Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπληρωθεί ακόμα περισσότερο από την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αντίσα Μπέμπα και ενισχύθηκε από την παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκεί. Μας δόθηκε η δυνατότητα να σας συναντήσουμε εκεί και να συναντήσετε κι εσείς πολλούς σημαντικούς ε, αντιπροσώπους οι οποίοι ε, είναι κατεστημένοι στην Αντίσα Μπέμπα και ασχοληθήκατε βέβαια ιδίω στην επίσκεψή σας του Σεπτεμβρίου με την καυτή επικαιρότητα και ιδίω με το ζήτημα της Λιβύης. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και όλες αποφάσισαν με την σημερινή συνεδρίαση να δώσουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο σε όλα αυτά τα ζητήματα και να καταφέρουμε να εντοπίσουμε τους τρόπους, τα μέσα με τα οποία θα καταφέρουμε να κινηθούμε μπροστά προκειμένου να υλοποιήσουμε τα διαφορετικά σημεία της στρατηγικής μας εταιρικής σχέσης. Θα ήθελα πολύ γρήγορα να φερθώ στο σημαντικότερο θέμα της ε, σημερινής συνεδρίασης, να αναφερθώ επίση στην ε, στρατηγική η οποία ισχύει προκειμένου να έχουμε ειρήνη, ασφάλεια και σταθεροποίηση πολιτική στην ε, Αφρική και να καταφέρω να αναφερθώ γρήγορα με τη δυνατότητα να επανέλθουμε εφόσον το επιθυμείτε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στις ε, προσδοκίες της Αφρικανικής Ένωσης ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πολύ μεγάλη αυτή προσπάθεια που καταβάλλεται προκειμένου να έχουμε μια Αφρική η οποία δεν θα διέπεται πλέον από κρίσεις και διενέξεις, αλλά μια Αφρική η οποία θα κινείται περισσότερο προς την ανάπτυξη και την ε, εμβάνθηση της διαδικασίας της δημοκρατικοποίησης και της ε, ολοκλήρωσης. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για την ε, συνεχή υποστήριξη που τα ευρωπαϊκά κράτη και συλλογικά και το καθένα ξεχωριστά έχουν ε, δώσει προς την ε, Αφρικανική Ένωση, καθώς επίσης και στις περιφερειακές οικονομικές κοινότητες, προκειμένου να προωθηθεί η ειρήνη στην Αφρική προκειμένου να σταθεροποιηθεί η δημοκρατική διαδικασία και να ενισχυθούν οι δυνατότητες των οργανισμών μας σε επίπεδο Αφρικανικής Υπήρου και σε περιφερειακό επίπεδο. Ως προς αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στην θετική εξέλιξη που έχουμε γενικότερα στο ζήτημα της ασφάλειας και της ειρήνης στην Αφρική. Σήμερα έχουμε πολύ λιγότερες συγκρούσεις στην Αφρική από ό,τι την προηγούμενη δεκαετία και έχουμε πολύ λιγότερα θύματα σήμερα από τις ένοπλες σειράξεις από ό,τι είχαμε την προηγούμενη δεκαετία. Καταφέρνουμε λοιπόν να εξηγιάνουμε περισσότερο την κατάσταση με τις διενέξεις. Έχουμε μία πρόοδο όσον αφορά την πρόληψη των συγκρούσεων και υπάρχει μια σαφής βούληση από πλευράς των κατοίκων της Αφρικής να υπάρχει μια ειρήνευση στις διάφορες συγκρούσεις και μια γενικότερη ε, βούληση για περισσότερη δημοκρατία, για περισσότερη ολοκλήρωση, για ενδυνάμωση των θεσμικών και ανθρωπίνων ικανοτήτων μας. Υπάρχει λοιπόν μια πραγματική δυναμική εξυγίανσης του γεωπολιτικού τοπίου, η οποία μάλιστα επιταχύνθηκε στην Αφρική, ιδίως ε, χάρη στην, ε, στο μετασχηματισμό του Οργανισμού της Αφρικανικής Ένωσης σε Αφρικανική Ένωση στις ε, αρχές του αιώνα αυτού, πριν από δέκα περίπου χρόνια προς όφελος όλων των ε, εταίρων, των συμμάχων που έχει η Αφρικανική Ήπειρος και που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια και ε, πρέπει να αναφερθώ βέβαια εδώ ότι ένας σημαντικός ε, σύμμαχος εταίρος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ξέρετε η Αφρική έχει πλέον πολλά και διαφορετικά μέσα η χρησιμοποίηση των οποίων μας επιτρέπει να διαδραματίσουμε σε Αφρικανική Ένωση ένα πρωταρχικό ρόλο στο ζήτημα της ειρήνης, της επίλυσης των συγκρούσεων και της ασφάλειας στην Αφρική. Έχουν γίνει λοιπόν, έχει γίνει εθαρρυντική πρόοδος, εκεί πέρα που παλιότερα τα πράγματα ήταν πολύ πιο ευάλωτα και εύθραυστα και έχουμε καταφέρει να διευθετήσουμε ε, διάφορες συγκρουσιακές ε, καταστάσεις και βλέπουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση σήμερα ότι ε, η διαδικασία επίλυσης των κρίσεων στις Κομόρες, στον Μπουρούντι, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στην ε, Κεντροφερκανική Δημοκρατία, στην ε, Γκουινέα Μπισάο. Σημειώνεται σημαντική πρόοδο σε όλες αυτές τις ε, περιοχές και χώρες και σιγά σιγά καταφέρνουμε να εξασφαλίσουμε την διέξοδο από την κρίση και την επίλυση των διενέξεων. Η Αφρικανική Ένωση προσπαθεί παράλληλα να συνεχίσει σε καθημερινή βάση όλες τις δραστηριότητές της σε όλους τους τομείς, όπως για παράδειγμα η διαφρομένη πρόληψη των συγκρούσεων, η επίλυση των συγκρούσεων, καθώς επίσης και η σταθεροποίηση και η εδραίωση της ειρήνης μέσω ενός φιλόδοξου προγράμματος για την ανοικοδόμηση, την αναδιάρθρωση μετά από περιόδους πολέμου. Η Αφρικανική Ένωση λοιπόν προσπαθεί να ενισχύσει κατά αυτόν τον τρόπο την Αφρικανική Αρχιτεκτονική Ειρήνης και Ασφάλειας που όπως το γνωρίζετε έχει ως βασικό της στοιχείο το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας το οποίο είχε πάνω από 300 συνεδριάσεις τελευταία χρόνια σε επίπεδο κρατών και κυβερνήσεων καθώς επίσης και σε επίπεδο υπουργών και μόνιμων αντιπροσώπων. Η Αφρικανική λοιπόν αρχιτεκτονική ειρήνη και ασφάλεια περισσότερο από ποτέ σήμερα διαρθρώνεται γύρω από την Αφρικανική δύναμη επιφυλακή με τις πέντε περιφερειακές ταξιαρχίες της και με τον υπηρετικό μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε επίσης και στην σημαντική πρόοδο που έχουμε σημειώσει όσον αφορά τις διάφορες δύσκολες καταστάσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια να τονίσουμε εδώ και τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλη αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει προκειμένου η αφρικανική αρχιτεκτονική ειρήνης και ασφάλειας να καταστεί πιο επιχειρησιακή. Η Αφρικανική Ένωση δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αναδιάρθρωση του θεσμικού της θεσμικής τάξης κάθε φορά που ε, προσπαθούμε να επέμβουμε σε χώρες όπου ε, υπήρξε στρατιωτικό πραξικόπημα. Πάλι με ιδιαίτερη ικανοποίηση μπορώ να πω ότι ε, η θεσμική αυτή τάξη πραγμάτων ειρηνικά κατάφερε να εδραιωθεί σε πολλές περιοχές προσπαθώντας να ξεπεράσουμε κάθε φορά τις εσωτερικές κρίσεις που υπήρχαν. Αναφέρομαι στην Μαυρετανία, στον Νίγηρα, καθώς επίσης και στην ιδιαίτερη περίπτωση της ακτής του Ελεφαντοστού. Πάλι βλέπουμε εδώ πέρα ότι η σταγματική τάξη επικράτησε. Στις αρχές του 2011 η διεθνής κοινότητα επικεντρώθηκε περισσότερο στην ε, υλοποίηση της γενικότερης ε, ε, συμφωνίας ειρήνης για το Σουδάν. Τώρα έχουμε την δημοκρατία του Σουδάν καθώς επίσης και τη δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν. Και εδώ καταφέραμε επίσης να έχουμε ένα δημοψήφισμα, του οποίου τα αποτελέσματα γίνανε δεκτά. Έχουμε λοιπόν ένα νέο κράτος, το κράτος του ε, Νοτίου Σουδάν, που ανήκει και αυτό με τη σειρά του στην Αφρικανική Ένωση και πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν ε, με την ε, γενικότερη συμφωνία ειρήνης, καθώς επίσης και με το συγκεκριμένο αυτό νέο κράτος, είναι ζητήματα τα οποία εξακολουθούν να μας απασχολούν. Υπάρχουν διάφορες χώρες όπως το Μπορούντι και η Νιγηρία που με τη συμμετοχή τους, με την καθημερινή τους δράση, συμμετέχουν στην θετική αυτή εμπειρία της δημιουργίας ενός νέου κράτους, του κράτους του Νοτιού Σουδάν. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι η Αφρικανική Ένωση είναι ιδιαίτερα δραστήρια όπως και τα Ηνωμένα Έθνη, με τα οποία ουσιαστικά έχει από κοινού την διαχείριση της Μινουάντ, καθώς της Ιουναμίντ, της υβριδικής αυτής αποστολής μεταξύ Αφρικανικής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών στον Ταρφούρ, έχει σημειωθεί και εκεί η πρόοδος προκειμένου να υποστηρίξουμε τη δυναμική των διαπραγματεύσεων, ιδίως στα πλαίσια της διαδικασίας της Ντόχα, με τη διευκόλυνση που έχουμε από το Κατάρ που ε, λειτουργεί ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στην Αφρικανική Ένωση και την Ηνωμένα Έθνη. Επίσης, ε, όσον αφορά τις ε, συνέπειες και όσον αφορά την προσοχή που πρέπει να δώσουμε, πρέπει να αφαιρθούμε και στο κέρας της Αφρικής, περιοχή η οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη, ασταθής, περιοχή επίσης η οποία βρίθει διαφόρων διαρθρωτικών ασταθειών και πρέπει να αφαιρθούμε εδώ πέρα πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση της Σομαλίας. Έχουμε μια αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στην Σομαλία, την Αμισόμ, και χάρη στην αποστολή αυτή οι ε, μεταβατικές διοικητικές αρχές κατάφεραν να κερδίσουν τον έλεγχο της πρωτεύουσας Αγκαμπισού και Κατάφεραν επίσης να απομακρύνουν διάφορες τρομοκρατικές ε, ομάδες από την ε, πρωτεύουσα την ε, Μογκαντισού. Ομάδες που με τη δραστηριότητά τους είχαν επηρεάσει πάρα πολύ την κατάσταση στην χώρα. Και βλέπετε ότι στη χώρα αυτή, στην Σομαλία, η δράση των οργανώσεων αυτών τρομοκρατικών ουσιαστικά έχει επηρεάσει ακόμα και την ανθρωπιστική βοήθεια, την προσπάθεια ανθρωπιστικής βοήθειας που γίνεται στην χώρα αυτή. Οι προσπάθειες που γίνονται σε περιφερειακό επίπεδο, στο κέρας Αφρικής, αλλά και σε γενικότερο επίπεδο της Αφρικανικής Υπήρου, αλλά και στο διεθνές επίπεδο, συμβάλλουν στο να ε, εδραιωθεί η ειρήνη, η ασφάλεια και σταθερότητα στη Σομαλία. Ο στόχος αυτός είναι πλέον υλοποιήσιμος και πιστεύω ότι θα πρέπει σε σχέση με αυτό να κινητοποιηθούμε περισσότερο. Επίσης, οι ε, δυνάμεις ε, της Κένια στην περιοχή της ε, Ζεμπόμ δημιούργησαν μια νέα κατάσταση. Βλέπουμε ότι η ομάδα Σαμπάμ έχει προχωρήσει σε μια αμυντική θέση. Διεξάγονται αυτή τη στιγμή διαβουλεύσεις προκειμένου να προσαρμοστεί η αποστολή Αμισόμ και χρειαζόμαστε και την διεθνή υποστήριξη, ιδίως των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποκριθούμε στην θετική αυτή εξέλιξη της επιτόπου κατάστασης. Θετική εξέλιξη που λογικά θα πρέπει να έχει ένα θετικό αντίκτυπο όσον αφορά τις πολιτικές προοπτικές της Σομαλίας καθώς επίσης και στην διαμόρφωση του ρόλου της διεθνούς κοινότητος στην χώρα αυτή. Τώρα, το ζήτημα του LRA αντιστασιακό στρατό του κυρίου είναι ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί και μας απασχολεί ιδιαίτερα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο ασχολήθηκε δύο φορές δύο συνεδριάσεις με το ζήτημα αυτό, με το ζήτημα του LRA. Και καταλαβαίνετε ότι ε, υπάρχουν πολλές ε, χώρες της Αφρικανικής Ένωσης και η ίδια η Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης που ασχολείται ιδιαίτερα με το ζήτημα αυτό. Υπάρχει μια πρωτοβουλία ενισχυμένης συνεργασίας, η οποία αποφασίστηκε υπό την αιγίδα της Αφρικανικής Ένωσης και η πρωτοβουλία αυτή βρίσκεται σε φάση υλοποίηση αυτή τη στιγμή με την έγκριση στι 22 Νοεμβρίου πριν από μερικέ μέρε από το Συμβούλιο Ασφάλεια και Ειρήνη Αφρικανική Ένωση, με ε, μιας ε, ενισχυμένης συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες της περιοχής εκείνης υπό την αιγύδα της Αφρικανικής Ένωσης και με την έντονη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ηνωμένων Εθνών και άλλων ε, διμερών εταίρων. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα τα οποία ανέφερα στην παρουσίασή μου δείχνουν τη γενικότερη θετική τάση που υπάρχει για την μείωση των συγκρούσεων και των διενέξεων στην Αφρικανική Ήπειρο και αυτό καταδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο σωστό δρόμο προς την εκπλήρωση της αποστολής της. Η εδραίωση όμως ε, της ειρήνης παραμένει ένα φιλόδοξο έργο και παραμένουν ακόμα διάφορα στάδια τα οποία πρέπει να βελτιώσουμε και πρέπει να συμπληρώσουμε. θα πρέπει να αποφύγουμε μια ειρηνευτική διαδικασία η οποία δεν θα έχει μια σταθερή βάση γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε άλλες διενέξεις πολλές φορές πιο βίες και πιο πολύπλοκες ακόμα. Έχοντας λοιπόν επίγνωση της κατάστασης αυτής η Αφρικανική Ένωση έχει ένα πλαίσιο δράσης για την αναδιάρθρωση και την οικοδόμηση μετά τις διενέξεις και για αυτό το λόγο συνεργάζεται με τις χώρες οι οποίες βγαίνουν από διενέξεις σε στενή συνεργασία με όλους τους εταίρους, αρχής γενομένης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να καταφέρουμε να εξαλείψουμε όλους τους ε, λόγους που οδηγούν σε κρίσεις και διενέξεις, που πολλές φορές συνδέονται με την ε, οικονομική και κοινωνική κατάσταση του πληθυσμού, καθώς επίσης και με το ζήτημα της διακυβέρνησης. Προκειμένου να ενισχυθεί περισσότερο ο διαθεσμικός μας διάλογος, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο πολύ λακωνικά αναφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως την Αραβική Άνοιξη. Πρόκειται για ένα μη ομοιόμορφο φαινόμενο εξελίξεων, το οποίο ουσιαστικά περνά από όλες τις φάσεις από όλες τις εποχές και όχι μόνο από την Άνοιξη, έχει πολλές διαφορετικές πτυχές, δεν παράγει παντού τα ίδια αποτελέσματα, αλλά αντίθετα υπάρχουν πολλά ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά για κάθε μία χώρα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, Αναφέρθηκα σε κάποια ζητήματα τα οποία θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας και είναι ζητήματα με τα οποία ασχολείται τόσο η Αφρικανική Ένωση όσο και οι ε, υπόλοιποι εταίροι μας, ζητήματα τα οποία αντιμετωπίσουμε με την πολύτιμη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. όλη αυτή η δράση μας, όλοι αυτοί οι τομείς δεν παρουσιάζουν την ε, ίδια πρόοδο. Η πρόοδος κάθε φορά εξαρτάται από τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών της Αφρικανικής Ένωσης, αλλά εξαρτάται και από τη συνεργασία που έχει η Αφρικανική Ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω για τι πολύ καλές σχέσεις και για την πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στην Αφρικανική Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως όσον αφορά την αρχιτεκτονική της ειρήνης και της ασφάλειας. Ολοκληρώνοντας, Χαίρομαι ιδιαίτερα για την δυνατότητα που μου δίνεται σήμερα να συμβάλλω κι εγώ στην εμβάθυνση του διαλόγου αυτού ανάμεσα στα θεσμικά μας όργανα και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Προτού συνεχίσουμε τη συζήτηση, θα δώσω το λόγο στον κύριο Westcott, που είναι Γενικός Διευθυντής για την Αφρική στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Κύριε Πρέσβη, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω στο ίδιο πάνελ, στην ίδια επιτροπή όπως μίλησε και ο εξοχότερος κύριος Πρέσβης. Ε, ο κύριος Επίτροπος ε, και θα αναφερθώ στα ίδια θέματα τα οποία προενέφερε εκείνος. Τα τρία βασικά θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή αφορούν ιδιαίτερα την Αφρική, την ειρήνη, την ευημερία και την συνεργασία. Ο κύριος επίτοπος μίλησε, αναφέρθηκε ιδιαίτερα για το θέμα της συνεργασίας και της ειρήνης και μιλάμε συνέχεια για τη μείωση του αριθμού των διαμαχών και των συγκρούσεων στην Αφρική, καταρχάς στο εθνικό επίπεδο, διότι οι περισσότερες συγκρούσεις που έχουν σημειωθεί στην Αφρική τα τελευταία 40-50 χρόνια δεν ήταν διαμάχες μεταξύ κρατών, αλλά εσωτερικές διαμάχες, εσωτερικές συγκρούσεις σε εθνικό επίπεδο. Οπότε ένα βασικό σημείο, ένα σημείο κλειδί του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να εδραιώσει υγιείς ε, θεσμικούς οργανισμούς, υγιείς θεσμούς για να μπορέσει να καταπολεμήσει τις ε, συγκρούσεις ε, και να βοηθήσει στην ειρήνευση. Αυτό βεβαίω ισχύει και σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο ολοκλήρου της Υπήρου της Αφρικής. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να οικοδομήσουμε αυτές τις, αυτούς τους θεσμούς, αυτά τα θεσμικά όργανα στις χώρες της Αφρικής. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητός ότι ο ρόλος μας σε μεμονωμένες χώρες είναι ε, ένας ρόλος ο οποίος εξελίσσεται ταυτόχρονα μέσα στις εσωτερικές προσπάθειες επίλυσης των συγκρούσεων. Σε περιφερειακό επίπεδο η ΕΚΟΒΟΣ, η ΕΚΟΒΑΣ, η ΣΑΝΤΕΚ, η ΙΚΑΤ ε, και άλλοι οργανισμοί έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην επίλυση διαφορών σε περιφερειακό επίπεδο και σε πολλές περιπτώσεις συγκρούσεων αυτοί οι περιφερειακοί οργανισμοί έχουν αναλάβει έχουν διαδραματίσει κέριο ρόλο ε, στον Ήγυρα, στην... Ε, Aims to play a supporting role. Στη Γουινέα. Uh, backing up. Ε, στην, ε, και κυρίως, επιβάλλοντας κυρίως ε, οικονομικές ε, κυρώσεις και άλλου είδους κυρώσεις από τους συναρμόδιους περιφερειακούς οργανισμούς. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με τη ΣΑΝΤΕΚ πολύ στενά για την επίλυση της πολιτικής κρίσης στη Μαδαγκασκάρη. και για την επίτευξη της συνταγματικής μεταρρύθμισης ε, στη χώρα αυτή. Συνεργαζόμαστε μαζί λοιπόν με τους περιφερειακούς οργανισμούς, αλλά και η Αφρικανική Ένωση συνεργάζεται με τους αφρικανικούς οργανισμούς και είμαστε πολύ ευτυχείς που η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι περιφερειακοί οργανισμοί συνυπέγραψαν ε, έναν οδικό χάρτη για την κατανομή των εργασιών που πρέπει να κάνει η κάθε πλευρά. Είμαστε Υποστηρίζουμε απολύτως την ε, προσέγγιση της επίλυσης των διαφορών από ε, αφρικανικές πηγές, από τους ε, τους ίδιους τους θεσμούς που ε, λειτουργούν στην Αφρική και είμαστε πρόθυμοι σε κάθε περίπτωση να συνυποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε τους οργανισμούς αυτούς στην επίλυση συγκρούσεων. Σας είπα λοιπόν, λειτουργούμε σε τρία επίπεδα, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν αυτών των ε, επιπέδων στην Αφρική πρέπει να συνεργαστεί στενά και με τον ΟΗΕ, με τη στο στην ακτή του Ελεφαντοστούν, ε, επίσης στην ε, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στο, με, την Άμισομ και την Γιούναμιτ στο, Σουδάν, Άμισομ στη Σομαλία, Γιούναμιτ στο Σουδάν ε, υπάρχουν ειδικοί εκπρόσωποι του ΟΗΕ οι οποίοι λειτουργούν σε αυτά τα μέρη και δρούν επιτόπου. Ε, προσπαθήσαμε να συγκεράσουμε σε ένα στρατηγικό πλαίσιο όλες τις ε, ενέργειες και τις επιχειρήσεις που πρέπει να γίνουν. Έχουμε αναπτύξει ένα στρατηγικό πλαίσιο για την περιοχή του Σαχέλ, με το, οποίο κυρίως άπτεται θεμάτων ασφάλειας της περιοχής και πριν από δύο εβδομάδες παρουσιάσουμε ένα παρόμοιο ε, πλαίσιο στρατηγικής για το κέρας της Αφρικής. Ε, αυτά τα στρατηγικά πλαίσια είναι πολύ σημαντικά για την εφαρμογή μέτρων που θα εδραιώσουν, θα αναπτύξουν ε, όλες τις προσπάθειες ειρήνης και ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ουσιαστικά το πλαίσιο ε, αφρικανικής ειρήνης και ασφάλειας και ιδιαίτερα ε, τον οργανισμό APF που είναι ο οργανισμός ε, ειρήνευση, αφρικανικής, υποστήριξης αφρικανικής ειρήνευσης, ειρήνευσης στην Αφρική. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε δύο οργανισμούς, η Άμισομ στην Σομαλία και η Μίκοπαξ, η οποία ε, προβλέπει την δημιουργία μιας αφρικανικής δύναμης για την κεντροαφρικανική δημοκρατία, στην, που θα λειτουργεί στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Οι δύο αυτές δυνάμεις, σε αυτές δύο έχουμε επενδύσει 240 εκατομμύρια ευρώ στην Άμισομ και στη Μήκοσιμ ε, για να ε, ξεκινήσουν τη λειτουργία τους. Είναι μια Αφρικανική πρωτοβουλία, είναι δύο δυνάμεις οι οποίες έχουν Αφρικανική ηγεσία ε, και η διαχείρισή τους γίνεται από την Αφρικανική Ένωση και τις εμπλεκόμενες δυνάμεις με τη βοήθεια του, των δυνάμεων ε, ασφαλείας του ΟΗΕ. Ε, εξετάζοντας ε, τώρα το μέλλον, των εξελίξεων στη Σομαλία, ο, Επίτροπος, ο κύριος Επίτροπε είπε ότι υπάρχουν ορισμένε ενθαρρυντικές ενδείξεις, αλλά απέχουμε πάρα πολύ από μια ολοκληρωμένη λύση. Εμείς στη Σομαλία υποστηρίζουμε ε, τρεις ενέργειες. Καταρχάς τις ενέργειες της Άμισομ. Ε, εδώ στα πλαίσια της Άμισομ μπορούμε να ενισχύσουμε τις δομές ώστε να είναι ασφαλείς. Δεύτερον, την TFG, ε, μέσω, και αυτό είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να προσφέρουμε εκπαίδευση, κατάρτιση ε, για τις ειρηνευτικές ε, ενέργειες που χρειάζονται για το πλαίσιο της ασφάλειας κλπ. Και τρίτον υποστηρίζουμε την όλη πολιτική διαδικασία μέσω του TFG συμπεριλαμβανομένης και της εξέβρισης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής, πολιτικής λύσης για την ε, διακυβέρνηση αυτής της χώρας για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι η χώρα αυτή θα έχει μια ισχυρή πολιτική, ένα ισχυρό πολιτικό μέλλον. Η Σομαλία λοιπόν είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς συνεργαζόμαστε, πώς οι διάφορες αυτές ε, ε, κλάδοι συνεργάζονται έτσι ώστε να επιτευχθεί κάποια πρόοδο στη Σομαλία αλλά πολλά περισσότερα πρέπει να γίνουν ειδικά φέτος. Έχουμε μία προθεσμία μέχρι τον Αύγουστο του 2012 για να ε, επιτύχουμε μία νέα συνταγματική διευθέτηση, μία νέα συνταγματική ρύθμιση. Σας συνεχίσουμε αυτή τη στιγμή να προσφέρουμε τη βοήθεια, να υποστηρίζουμε την άμυσο, αλλά θα δούμε μήπως χρειάζονται ε, άλλοι, ε, ε, άλλες πτυχές ενίσχυσης και βοήθειας, με ποιους άλλους τρόπους μπορούμε να βοηθήσουμε. Μέσω του APF επίσης και με την Αφρικανική Ένωση υποστηρίζουμε διάφορους εκπαιδευτικούς φορείς που δίνουν τη δυνατότητα στις αφρικανικές δυνάμεις να ενεργούν σε αποστολές ειρήνευσης και ασφάλειας, κυρίως στην Ανατολική Αφρική. Υπάρχει και στην Γκάνα το, το κέντρο ειρήνης ε, Κόφιανάν, του ίδρυσε Κόφιανάν. Επίσης, ε, υπάρχει ένα άλλο κέντρο, Αμάνι Αφρικα λέγεται, όπου προσπαθούμε να προσφέρουμε κατάρτιση και εκπαίδευση στις ε, δυνάμεις, στις έκτακτες ε, δυνάμεις, στις δυνάμεις επιφυλακής. Και τρίτον, υποστηρίζουμε τη διαχείριση κρίσης, ΣΥΤΣΕΝ, στα πλαίσια της Αφρικανικής Ένωσης για την πρόληψη των συγκρούσεων και κρίσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν διαμέσου της Αφρικανικής Ένωσης προσφέρει και ενεργεί μέσω διαφόρων ε, οδών και καναλιών. Επίσης στη Λαϊκή Δημοκρατία Δημοκρατία, στη Δημοκρατία του Κονγκό αυτή τη στιγμή έχουμε προσφέρει τη βοήθειά μας για τις εκλογές, τις τρέχουσες εκλογές που γίνονται και επίσης μια ισχυρή στατιωτική και αστυνομική δύναμη στην ε, ε, Δημοκρατία του Κονγκό και έχουμε επίσης ε, βοηθήσει πάρα πολύ σε ενέργειες ελέγχου πλήθους. πλήθους. διαδηλώσεων, διαταραχών κλπ. Και εξετάζουμε συγκεκριμένα μέτρα αυτή τη στιγμή για να ενισχύσουμε τις ενέργειες κατά πολέμησης της θαλάσσιας πειρατείας, αναπτύσσοντας μία παράκτια δύναμη, ε, εν είδη ακτοφυλακής δηλαδή, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα το μεγάλο θέμα αυτό της πειρατείας. Τώρα πάλι λίγο ανισχυτική είναι η κατάσταση στο Σουδάν όπου χρειαζόμαστε να πρέπει να συνεργαστούμε πολύ στενά με την Αφρικανική Ένωση και με την Ίγκαρτ για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα εκεί έχουμε υποστηρίξει τις διπλωματικές ενέργειες του Προέδρου Μπέκη της Νοτιού Αφρικής Έχουμε επίσης και κρυμείς υποθέσεις στα πλαίσια της CPA. Είναι μια πάρα πολύ ευάλωτη, ευαίσθητη και δύσκολη κατάσταση ε, και στο Σουδάν και πρέπει να συνεργαστούμε πολύ στενά όχι μόνο με τον πρόεδρο Μπέκη αλλά και με τον ΟΗΕ και με την Αφρικανική Ένωση. Ε, αυτή τη συνεργασία την επιτελούμε διαμέσου του εκπροσώπου μας της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας έδωσα λοιπόν μια σύντομη επισκόπηση όλων των ε, ενεργειών μας και των οργανισμών διαμέσου των οποίων λειτουργούμε. Ε, ευχαριστώ κύριε Γενικέ. Προτού δώσω το λόγο στους συναδέλφους που θέλουν να πάρουν το λόγο, θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα στον ε, κύριο Πέσβη Λαμάμρα. Πρώτον, σχετικά με την αφρικανική δύναμη επιφυλακής που παραμένει μια ε, δύναμη η οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν και είναι μια φιλόδοξη δύναμη. Πώς το βλέπετε, ε, η υλοποίησή της έχει μετατεθεί μέχρι το 2015. Ο στρατηγός ε, από την Κινέα θα έχει αναλάβει τις τα καθηκόντά του. Πώς βλέπετε την δομή της, ποια, τι είδους συγκεκριμένη συνεργασία θα αναμένατε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τομέα. Δεύτερο, για τη Σομαλία έχετε αναφερθεί εκτενώς στο θέμα της σύγκρουσης αυτής. Μας μιλήσατε και για τις στρατιωτικές ε, πρόοδους που έχουν γίνει με την ε, δύναμη Αμισόμ. Έχουμε μεταβεί ε, στην Ουγκάντα. Πήγαμε την Άνοιξη. Είχαμε μια εις ανταλλαγή απόψεων με τους, τις αρχές της Ουγγάντας, ήταν και ο αντιπρόεδρος Πάσκου και μας ε, εντυπωσίασε βέβαια η δέσμευση της Ουγγάντας και από το αίτημα της Ουγγάντας και του Μπουρούντι, το συνεχόμενο, για τη διεύρυνση ε, της ε, Αμισόμ και της συνεισφοράς του σε άλλες αφρικανικές χώρες πού βρισκόμαστε σε αυτό το θέμα. Τα αιτήματα τη Ουκάντα και του Μπουρούντι επανέρχονται. Ποιες είναι οι απαντήσεις που μπορεί να δώσει η Αφρικανική Ένωση δεδομένης της εξέλιξης ε, της κατάστασης του Μογκαντήσου ε, μπορεί τα πράγματα να μην είναι τόσο έντονα όσο ήταν όταν μεταβήκαμε εμείς τότε. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου, ο κ. Γκάλερ ο οποίος είναι ο συντονιστής του ΕΛΚ. Θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά και μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διερμηνία βεβαίω στις γλώσσε σα. Yeah. Okay. Yeah, um, Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον ε, πρέσβη και επίτροπο της Αφρικανικής Ένωσης, κύριο Λαμάμρα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι εδώ μετά από την επίσκεψή μας στην Αντισάμπεμπα, λίγο μετά την επίσκεψή μας σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ε, προθυμία που δείχνετε και τη δέσμευση που έχετε αναλάβει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυσης της συνεργασίας. Αυτή η συνεργασία μας ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής είναι μία από τις πιο δραστήριες ένα από τα πιο επιτυχημένα και δραστήρια πλαίσια συνεργασίας μέχρι σήμερα. Και πιστεύω και στο μέλλον να εξελιχθεί, να ακολουθεί στην ίδια πορεία Ήδη αναφέρεται πολλές προβληματικές περιοχές, πολλούς προβληματικούς τομείς. Συζήτησα με πολλούς συναδέλφους στην τελευταία κοινοβουλευτική συνεδρίαση που έγινε την περσμένη εβδομάδα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών και και μου επιβεβαίωσαν τα μεγάλα προβλήματα και στην περιοχή του, Σαχέλ και στην περιοχή της Σομαλίας. Έχω λοιπόν καταρχάς μία ερώτηση. Από ό,τι φαίνεται η Αλ Σαμπάχ, η παραστατιωτική οργάνωση Αλ Σαμπάχ στη Σομαλία έχει αποδυναμωθεί διότι οι οικονομικοί πόροι που μέχρι τώρα προέρχονται από τη Λιβύη έχουν στερέψει και μέχρι τώρα Έχουμε την εντύπωση ότι στις δυσκολίες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κάποια αλλαγή στην τακτική που εφαρμόζει η Al-Shabaab διότι δεν μπορεί να πληρώσει πλέον. Δεν μπορεί να πληρώσει τα μέλη της και έτσι ψάχνουν να βρουν ε, μια διαφορετική προπαγάνδα, παραδείγματο χάρη τον εθνικισμό, χρησιμοποιούν εθνικιστική, ε, εθνικιστικά συνθήματα εναντίον όλων των εξωτερικών εχθρών, παραδείγματο χάρη της Κένιας. Και θα ήθελα να ρωτήσω, ε, εάν θα ήταν πολιτικά, πολιτικά ενδεδειγμένο να ενισχύσουμε τις εντολές της Άμισομ για να συμπεριλάβουμε εκτός των ειρηνευτικών ενεργειών και τη δυνατότητα ενίσχυσης και δυνάμεων και ενδεχομένως στο μέλλον και σομαλικών δυνάμεων, έτσι ώστε να μπορούν να στραφούν κατά της αλ ε, και να καταπολεμήσουν αυτά τα εθνικιστικά τις εθνικιστικές φωτιές τις οποίες ανάβει τώρα η αλ ε, είναι μια ερώτηση αυτή που απευθύνεται και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αν αυτό είναι κάτι το επισημητό. Δηλαδή βλέπετε τη δυνατότητα αυτή την εντολή της Άμισομ να την αναθεωρήσουμε, να την εμπλουτίσουμε αν θέλετε έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει και ενέργειες ε, στοχειωτικών δυνάμιο της Κένιας ή και της Σομαλίας ας πούμε για την ε, διασυνοριακή συνεργασία, ένοπλη συνεργασία. Ίσως θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο επιτέλους να, να λήξει αυτή η ιστορία με την Αλ-Σαμπάχ στη Σομαλία. Όσον αφορά την κατάσταση στο Σαχέλ, ιδιαίτερα από τη Μαυριτανία, Μαλή, τον Ήγηρα, το Τσάντ, οι συνάδελφοι μας είπαν ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό μετά την απόσυρση των ε, ειρηνευτικών δυνάμεων και ότι αυτή τη στιγμή οι διάφορες ένοπλες ομάδες εκεί ε, προμηθεύονται όπλα, μεγάλες ποσότητες ε, όπλων ε, και εξοπλισμού, στρατιωτικού εξοπλισμού και αυτό ανησυχεί ιδιαίτερα τις γειτονικές χώρες, το Μαλί και άλλες, διότι υπάρχει αυτό το κενό, το κενό πλέον εξουσίας και έτσι αυτές οι ομάδες μπορούν ελεύθερα να προγραμματίσουν τις ενέργειές τους, να αγοράσουν άλλα όπλα, να αποθηκεύσουν τα όπλα τους για να προγραμματίσουμε την ησυχία τους εν συνεχεία ένοπλες συγκρούσεις στο μέλλον. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανησυχία ότι αυτές όλες οι δυνάμεις έχουν πολύ στενές σχέσεις με την Αλκαΐντα. Τι νομίζετε λοιπόν ότι μπορεί να γίνει για να δημιουργηθεί μία κυρίαρχη ε, εδαφική επικράτεια, ε, ελεύθερη εδαφική επικράτεια, αλλά να έχει μία κυρίαρχη βάση αυτή η επικράτεια, σε να μην υπάρχει κενό εξουσίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκουαλτιέρη, που είναι συντονιστής των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ τον πρέσβη Λαμάμπρα. Το πρώτο που θα ήθελα να κάνω είναι να συμφωνήσω με τον Γενικό Διευθυντή και με τον κύριο Γκάλερ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε εδώ και τονίσατε πόσο σημαντική είναι αυτή η συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρικανική Ένωση. Ιδιαίτερα αυτή την συνεργασία για την ασφάλεια και την ειρήνη. Έχω μία ερώτηση την οποία θα ήθελα να απευθύνω στον πρέσβη αλλά ε, μέσα από τις ερωτήσεις του κ. Γκάλερ και του Νταν έχουμε ήδη ακούσει τα θέματα αυτά, ιδιαίτερα για την κατάσταση στην Σομαλία. Έχουμε λάβει μια σειρά από ειδήσει από την περιοχή αυτή και έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα, ακόμη και αν δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα τα ζητήματα. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα μεταβαλλόμενα σενάρια ε, στην ε, θητεία και στην εντολή αυτής της αποστολής για την ειρήνη και την ασφάλεια και επίσης σχετικά με τον άμεσο ρόλο της Άμισομ τι στήριξη θα μπορούσαμε να προσφέρουμε και εσείς τι στήριξη θα μπορούσατε να προσφέρετε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι ρόλο διαβλέπετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο μας. Ε, τι σημεία θα πρέπει να ξαναδούμε επιγόντως σε αυτό το θέμα. Και γενικώ ομιλούντες τώρα στο θέμα του Ταμείου για την Ειρήνη στην Αφρική. Είναι μια ερώτηση που απευθύνεται κυρίως προς τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Westcott Η συνεργασία που έχουμε είναι πολύ γερή σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά τους πόρους, τις δομές ε, που θα ε, ε, χρησιμοποιηθούν. Και φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα τα οποία πρέπει να τύχουν διαχείρισης για την χρήση των διαθροτικών ταμείων. Αλλά ε, με την χρήση άλλων ταμείων και πόρων. Αυτό θα ήταν μία επιλογή για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα ε, της, του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαμε να έχουμε το Ταμείο για τη Σταθερότητα. Υπάρχουν κάποια κονδύλια για την ασφάλεια. Η ερώτηση λοιπόν είναι από την προοπτική του Κοινοβουλίου, δεδομένης της σημαντικότητας αυτής της συνεισφοράς και της, ε, σε μεγάλη κλίμακα χρήσεως ε, των ταμείων αυτών μαζί με τους Αφρικανούς συναδέλφους. Σε ποιο βαθμό θα μπορούσε το Ευρωκοινοβούλιο να βοηθήσει στον προσδιορισμό μιας πολιτικής ασφάλειας, που να μην είναι απλά μια αναπτυξιακή πολιτική. Πώς θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε ότι η πολιτική ασφάλειας συμβαδίζει με την αξιολόγηση της κατάστασης, ιδιαίτερα της ε, τις σχέσεις κόστους και ωφέλειας. Γιατί ε, μου φαίνεται ότι αυτό το πολιτικό πλαίσιο θα πρέπει να γίνει αποτελεσματικό. Ε, θα πρέπει να είναι πολύ αποτελεσματικό. Δεν ήταν μέχρι στιγμής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας συγχαρώ για ε, αυτά που παραθέσατε εδώ, το θέμα της συνεργασίας ανάμεσα στην Αφρική και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει πολύ σημαντικό και για τα δύο, τις δύο περιοχές, και την Αφρική και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω ερωτήσεις που σχετίζονται με το θέμα της ασφάλειας και της κατάστασης ασφάλειας στην Αφρική διότι σε διάφορες περιοχές η κατάσταση της ασφάλειας παραμένει πολύ ανησυχητική. Η Σομαλία είναι μια μεγάλη ανησυχία για μας ε, λόγω των πειρατών, γιατί οι οικονομικές ζημίες είναι μεγάλες και για την Ευρώπη και για σας. Αλλά ε, ανησυχώ ότι αν, κατά πόσο το κράτος της Σομαλίας έχει τη δυνατότητα να, να αντεπεξέλθει και να αντιδράσει. Και πιστεύω ότι στην ε, περιφέρεια αυτή υπάρχει μια πραγματική τάση διαχωρισμού. Είχα την δυνατότητα να μιλήσω με εκπροσώπους από τη Σομαλία και πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν αυτή την οδό Δηλαδή θα προσπαθήσουν να χωρίσουν τις περιφέρειες ως ε, ξεχωριστά κράτη. Είναι ένας κατακαιρματισμός που παρατηρείται στην Αφρική. Εάν ε, δούμε τι συνέβη και στο Σουδάν, για παράδειγμα. Ε, λόγω του δημοψηφίσματος, τα δύο κράτη συνέχισαν να έχουν προβλήματα. Πώς βλέπετε αυτή την τάση κατακαιρματισμού, εδαφικού κατακαιρματισμού της περιφέρειας και τι άποψη έχετε σχετικά με τις ε, προσπάθειες της δικές σας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον μετριασμό ε, του αντικτύπου των ε, πειρατιών έχουμε ένα ε, άλλο σημαντικό πρόβλημα, γιατί όπως έχει ήδη διαπιστωθεί, δεν υπάρχουν σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα της δικαιοσύνης. Τι μπορούμε να κάνουμε στο θέμα αυτό, διότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα του καθενός να προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Ε, πιστεύω ότι αυτοί που εμπλέκονται στην πειρατεία έχουν την τάση να συνεχίζουν, διότι η αντίδραση της Αφρικανικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι αρκετά έντονη στο θέμα αυτό. Όταν είχα μεταβεί στο Τζιπουτί και είχα μιλήσει με τους εκπροσώπους μας, ε, ε, άκουσα ε, για την ανάγκη να υπάρχει μια επέκταση της θητείας της δύναμης εκεί και θεωρούν ότι η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ δεν τους επιτρέπει να έχουν ισχυρή αντίδραση και αντίκτυπο στην περιοχή. Δύο θέματα λοιπόν, δύο ερωτήσεις αυτές. Η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με την Αραβική Άνοιξη. Ε, αυτή η προσέγγιση βιβάλτη τύπου τεσσάρων εποχών ε, πιστεύω ότι τα αποτελέσματα της Αραβικής Άνοιξης θα επηρεάσουν τη συνεργασία ανάμεσα στην Αφρική Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ξέρετε, στην διάσκεψη κορυφής της Τρίπολης ε, καθορίστηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές συνεργασίας ανάμεσα στις, στα δύο όργανα, στις δύο και αρχίσαμε ήδη να κάνουμε κάποια πράγματα. Αλλά εσείς πιστεύετε ότι η εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης στη Βόρεια Αφρική θα επηρεάσει τους κανόνες συνεργασίας ανάμεσά μας ή μήπως θα δημιουργήσει άλλες προτεραιότητες στη συνεργασία μας. Σας ευχαριστώ. Merci, Monsieur Στάτσνικ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος γιατί βλέπετε η Αφρική είναι μια τεράστια ήπειρο, επομένω προκύπτουν πάρα πολλά ερωτήματα, πάρα πολλές ζώνε ενδιαφέροντο υπάρχουν. Θα ήθελα να απευθυνθώ και στου δύο μιλητέ μα και να του ζητήσω να μιλήσουν λίγο περισσότερο για το πώ έχουν τα πράγματα στο Νότιο Σουδάν καθώ επίση και στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Είμαστε ικανοποιημένοι με την υφιστάμενη κατάσταση και είστε αισιόδοξοι για το προσεχέ μέλλον. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Κύριε Πρέσβη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω τα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έθεσαν πολύ σημαντικά ερωτήματα, πολύ κέρια ερωτήματα. Να ξεκινήσουμε τα δικά σας κύριε Πρόεδρε. Η δύναμη επιφυλακής. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα σχέδιο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, σε φάση υλοποίησης. βέβαια η ταχύτητα με την οποία οι διάφορες συνιστώσεις της ε, δύναμης αυτής αναπτύσσονται εξαρτάται από πολλές ε, και διάφορες προϋποθέσεις και μπορεί προφανώς να επηρεάσει με τον έναν τρόπο τη δυνατότητα αποτελεσματικότητα. Σας είπαμε ότι έχουμε πέντε ταξιαρχίες σε διάφορες γεωγραφικές ζώνες της Αφρικανικής Υπήρη. Έχουμε τρεις ε, ταξιαρχίες που έχουν ήδη συμπληρώσει όλες τις ασκήσεις που έπρεπε να λάβουν χώρα προκειμένου να πιστοποιηθεί η δυνατότητά τους να συμμετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές. Οι δύο εναπομείναντες ταξιαρχίες έχουν κάποια καθυστέρηση όσον αφορά τη συμπλήρωση αυτών των ασκήσεων. Μπορέσαμε να κάνουμε σε επίπεδο Αφρικανικής Υπήρου μια άσκηση στρατιωτικής διοίκησης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στέφθη με επιτυχία στην δεύτερη άσκηση που ξεκίνησε στην Αντίσα Μπέμπα πριν από μερικές εβδομάδες. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια άσκηση που θα συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις ταξιαρχίες, τρεις από τις πέντε, και θα έχουμε μια προσωμείωση πραγματικής στρατιωτικής ανάπτυξης. Προφανώς υπάρχουν κάποιες προκλήσεις τις οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε, κάποια προβλήματα στρατηγικής κινητικότητας πρέπει πολλές φορές να έχουμε τη δυνατότητα για θαλάσσιες και αεροπορικές ε, μεταφορές. Έχουμε την πρόκληση επίσης της χρηματοδότησης, υπάρχουν κάποιες δημοσιονομικές στενότητες. Έχουμε επίσης την πρόκληση της ε, τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης, προκειμένου να υπάρχει η απαραίτητη διασύνδεση ανάμεσα στις μάχημες μονάδες. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα, προκλήσεις, τα οποία προσπαθούμε πολύ ενεργά να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε επίσης ε, τακτικές συναντήσεις των επικεφαλής ΓΕΘΑ καθώς επίσης και των Υπουργών Άμυνας των ε, κρατών μελών της Αφρικανικής Ένωσης και χάρη στις συναντήσεις αυτές καταφέρνουμε επίσης να συντονίσουμε καλύτερα τη δραστηριότητα της δύναμης επιφυλακής και καταφέρνουμε να κάνουμε και ένα καλύτερο προγραμματισμό για τα επόμενα έτη. Θεωρούμε πάντως ότι η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα επικοδομητική. Στην τελευταία μας συνάντηση των Υπουργών Αμήνης και των Επικεφαλής των Στρατικών Δυνάμεων αποφασίσαμε σε κάθε μία από τις ταξιαρχίες αυτές να έχουμε και μία ναυτική ικανότητα, ναυτική δύναμη προκειμένου να καταπολεμήσουμε την πειρατεία κάθε μία ταξιαρχία να είναι σε θέση δηλαδή να καταπολεμά την, τα φαινόμενα πειρατείας και προκειμένου να καταφέρουν οι ταξιαρχίες αυτές να διεξάγουν και κάποιες περιπολίες περιβαλλοντικής προστασίας, ιδίως όσον αφορά διάφορα τοξικά απόβλητα στις α, θάλασσες και για να καταφέρουν να καταπολεμήσουν και άλλα φαινόμενα όπως η διακίνηση ναρκωτικών. Επομένως η ε, ναυτική αυτή συνιστόσα αποτελεί ένα νέο στοιχείο, ένα νέο χαρακτηριστικό των ταξιαρχιών αυτών της δύναμης επιφυλακής που θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε καλύτερα σε διάφορες προκλήσεις που καλείται τώρα να αντιμετωπίσει η Αφρική και για τις οποίες δεν είχε τα απαραίτητα μέσα αντιμετώπισης στο παρελθόν. Ο πρώην Υπουργός Αμήνης, ε, στρατηγός ε, Γκούνταμπε είναι ο επικεφαλής της ε, αφρικανικής δύναμης αυτής επιφυλακής εδώ και ένα χρόνο και πιστεύω ότι ε, προσφέρει ουσιαστικά μια πολύ σημαντική τεχνογνωσία στις νέες του αυτές αρμοδιότητες αλλά και σε πολιτικό επίπεδο η παρουσία του στρατηγού Κονατέ στην ε, γενικότερη αρχιτεκτονική δομή της Αφρικανικής Ένωσης ε, καταδεικνύει την ε, δημοκρατική μετάβαση που πλέον χαρακτηρίζει πάρα πολλές χώρες ε, στην Αφρικανική Ένωση. Επίσης, όσον αφορά την Αφρικανική δύναμη επιφυλακής, θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμα. Πέρα από τις στρατιωτικές επιχειρησιακές ιδιαιτερότητές της, η Αφρικανική δύναμη επιφυλακής αποτελεί ουσιαστικά ένα μέσο επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων στην Αφρική. Στο παρελθόν υπήρχαν ε, πολλές διαφορετικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Αφρική. Θα θυμάστε ότι είχαμε πάρα πολλά προβλήματα συνοριακής φύσης ανάμεσα σε όμορες χώρες. Έπρεπε πλέον να καταφέρουμε να έχουμε μία κοινή προσέγγιση όσον αφορά την στρατιωτική δύναμη στην Αφρική. Στο παρελθόν αντιμετωπίζαμε πολύ συχνά τις όμορες χώρες ως εχθρικές χώρες. Τώρα οι όμορες, οι γειτονικέ χώρες αποτελούν στρατιωτικό σύμμαχο για την αντιμετώπιση διάφορων φαινομένων όπως φυσικές καταστροφές ή εξωτερική κίνδυνη. Αντιμετώπιση φαινομένων όπως η πειρατεία για παράδειγμα. Και η η συνεργασία αυτή μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να προασπιζόμαστε τα θεσμικά όργανα των δημοκρατιών μας και καταφέρνουμε να έχουμε πλέον μια κοινή προσέγγιση, μια κοινή έννοια όσον αφορά την ασφάλεια και την ειρήνη στην Ήπειρο. Η διάσταση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, δεν την υπογραμμίζουμε αρκετά συχνά, πάντως ήθελα να την τονίσω ιδιαίτερως σήμερα στη σημερινή μας συζήτηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο δικός χάρτης υπαριθμών 3, ο οποίος εγκρίθηκε από τους υπουργού αμήνης στη συνεδρίαση που είχαμε τον Οκτώβριο, έχει ως στόχο να θέσει σε πλήρη επιχειρησιακή φάση την Αφρικανική Δύναμη Φυλακή το 2015. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουν επιληθεί, ότι θα έχουν διευθετηθεί όλα τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον τρει από τις πέντε ταξιαρχίες θα είναι σε θέση να εμπλακούν σε επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης και αυτό από μόνο το αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Πρέπει να σας πω ότι στο εσωτερικό κάθε μιας, κάθε μιας από αυτές τις ταξιαρχίες υπάρχει και μια ομάδα α, ταχείας ανάπτυξης, πράγμα το οποίο μας επιτρέπει να επεμβαίνουμε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα ταχύτατα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η θέση σε επιχειρησιακή φάση ουσιαστικά τι σημαίνει. Σημαίνει να καταφέρνουμε να επεμβαίνουμε ε, γρήγορα, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, κάθε φορά που καλούμαστε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτές ε, οι μονάδες ταχείας ανάπτυξης στα πλαίσια της αφρικανικής δύναμης επιφυλακής θα μας ε, επιτρέψουν να καταφέρουμε να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο το σημαντικό αυτό εγχείρημα. Όσον αφορά τώρα τη Σομαλία, πολλοί ομιλητέ αναφέρθηκαν στη χώρα αυτή, απαντώντας πιστεύω σε όλα τα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν για τη Σομαλία, θα ήθελα να πω καταρχάς ότι ε, αναμφισβήτητα η Σομαλία αποτελεί πολύ σημαντική πρόκληση για την Αφρική, μια πολύ σημαντική πρόκληση την οποία όμως μοιράζεται η Αφρικανική Ένωση με την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα. Για 20 χρόνια δεν είχε κυβέρνηση η χώρα αυτή και για 20 χρόνια η Σομαλία αποτελούσε κίνδυνο όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για την ίδια και κατάφερε να γίνει βέβαια και κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία μέσω των φαινομένων πειρατείας και μέσω του, των φαινομένων διεθνούς τρομοκρατίας απειλεί πλέον και τη διεθνή ασφάλεια. Είναι πλέον σαφές ότι η ομάδα Al-Shabaab συνδέεται με την Al-Qaeda. Επομένως, ε, ο αγώνας που δίνεται για τη σταθεροποίηση της Σομαλίας είναι ένας αγώνας για την ίδια τη δημοκρατία στη Σομαλία, για τη συμφιλίωση των Σομαλών, για τις καλές συνθήκες γειτονίας στο κέρας Αφρικής, αλλά και ένας αγώνας ο οποίος δίδεται για τα επικίνδυνα αυτά φαινόμενα, την πειρατεία δηλαδή και τη διεθνή τρομοκρατία. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν σφαιρικά το ζήτημα της Σομαλίας, είναι σαφές ότι ε, όλα τα όσα γίνονται, όλες οι επενδύσεις που λαμβάνουν χώρα, δυστυχώς ξεκινώντας από το αίμα το οποίο χύνουνε ή χύνεται από τους γενναίους στρατιώτες, τόσο της Σομαλίας όσο και του Μπουρούντι, προσπάθειες οι οποίες γίνονται όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την αποστολή της, της Αμισόμ. 25.000 ήταν οι στρατιώτες που τα τελευταία χρόνια συμμετείχαν στα πλαίσια της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών. Βλέπουμε τώρα ότι έχουμε μία αποστολή, την Αμισόμη, η οποία ξεκίνησε έχοντας κάποια πολύ στοιχειώδη στοιχεία και έφτασε περίπου τους 9.800 στρατιώτες με ανώτιτο πλαφόν τους 12.000. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ε, πολλοί παράγοντες που επηρέασαν την εξέλιξη της κατάστασης και σήμερα έχουμε βρεθεί πλέον με ένα σαφές όραμα όσον αφορά την πολιτική κατάσταση της Σομαλίας και έχουμε και κάποιες επιτόπου προοπτικές οι οποίες είναι σαφώς υλοποιήσιμες και είναι ρεαλιστικές και υπάρχει μια συνεργασία ανάμεσα στην πολιτική και την στρατιωτική πτυχή της δράσης μας και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε πριν τις 20 Αυγούστου του 2012 θα είμαστε λογικά σε θέση να έχουμε ένα νέο σύνταγμα στη Σομαλία, να έχουμε φαινόμενα συμφιλίωσης και εκδημοκρατισμού, θα έχουμε δράση προκειμένου η παραστρατιωτικές ε, ένοπλες οργανώσεις να έχουν ταχθεί υπό την ε, μεταβατική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Συμφωνώ επίσης ότι η ομάδα Al-Shabaab έχει εξασθενήσει, αλλά θα πρέπει ουσιαστικά οι ε, ένοπλοι αυτοί νέοι που συμμετέχουν στην Al-Shabaab και οι οποίοι ουσιαστικά ψάχναν εργασία και δεν κατάφεραν να την αποκτήσουν με νόμους τρόπους, απευθύνθηκαν πολύ συχνά στην τρομοκρατική αυτή οργάνωση που πληρώνει ουσιαστικά τους νέους στους οποίους στρατολογεί πολύ περισσότερο από ό,τι θα μπορούσε να τους πληρώσει ποτέ η μεταβατική κυβέρνηση της χώρας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει και μια έντονη οικονομική πτυχή στο όλο πρόβλημα, πέρα από τον φανατισμό, του πολύ σκληρού πυρήνα της αλ shabaab Και αυτό βέβαια ισχύει και προφανώς οι άνθρωποι αυτοί, οι πιο εξτρεμιστές, συνδέονται με την Αλκάιντα και συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση που έκανε ο κύριο Γκάλερ. Προφανώς στα πλαίσια της Αλ-Σαμπάμπ υπάρχει μία τάση διεθνοποίηση μεγαλύτερης διασύνδεσης με την Αλκάιντα Υπάρχουν διάφορε ομάδε ε, σε εθνικό επίπεδο που έχουν προσπαθήσει προφανώ να αναλάβουν ακόμα και την ε, εξουσία. Και καταλαβαίνετε ότι ε, αυτό πολλές φορές δημιουργεί συγκρούσεις ανάμεσα στις διάφορες ένοπλες ομάδες της χώρας. Όσον αφορά την Al-Shabaab, έχουν χάσει τον έλεγχο της βασικής αγοράς της Μογκαντισού αυτή τη στιγμή ε, η Αμισόπιμα, καθώς επίσης και οι δυνάμεις της μεταβατικής κυβέρνησης κατάφεραν να εξαλείψουν την Αλ-Σαμπάμπ από την Μογκαντισού, προφανώς έχουμε οδηγηθεί σε μια εξασθένηση της ομάδας αυτής. Επίσης είναι σαφές ότι υπάρχουν ε, διάφορες πηγές ε, χρηματοδότησης, κρατικές, παρακρατικές και άλλες, τις οποίες προφανώς πρέπει να εξαλείψουμε. Όσον αφορά τώρα την εντολή, την θητεία της Αμισόμα, πρέπει να σας πω ότι δόγμα της Αφρικανικής Ένωσης είναι η υποστήριξη της ειρήνης και όχι peacekeeping, υποστήριξη της ειρήνης. Τι σημαίνει υποστήριξη της ειρήνης. Σημαίνει ότι η Αφρικανική Ένωση μπορεί ουσιαστικά να συμμετέχει, να παρεμβαίνει στις περιοχές εκείνες όπου δεν υπάρχουν δυνάμεις του ΟΗΕ οι οποίες έχουν ως στόχο να συναυθεί μια συμφωνία ειρήνης. Έχουμε διάφορες αποστολές όπως η ΑΜΗ στον Ταρφούρ το 2004, αποστολή η οποία είχε εδραιωθεί εκτός οποιασδήποτε συμφωνίας ειρηνευτικής και η ΑΜΙΣΟΠ ξεκίνησε προτού καν αρχίσει η διαδικασία του Τζιμπουτί που οδήγησε στη συμφωνία τελικά του Τζιμπουτί που ήταν προφανώς μια συμφωνία κυβερνητική. Ακολουθούμε λοιπόν αυτή τη διπλωματική έννοια της υποστήριξης της ειρήνης και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση τελικά όπου η Αμισόμ έχει εξουσίες αρμοδιότητες ε, υλοποίησης της ειρήνης μέσω της ε, ε, προσφυγής της, στη χρησιμοποίηση στρατιωτικής δύναμης. Καλούμαστε δηλαδή να αναλάβουμε την απαραίτητη δράση προκειμένου να προστατεύσουμε τα νέα θεσμικά όργανα της μεταβατικής κυβέρνησης. Αν η λοιπόν δεν είχε καταβάλει σημαντικές προσπάθειες και αν δεν είχε συνταχθεί τελικά με τις δυνάμεις της μεταβατικής κυβέρνησης για την απελευθέρωση της πρωτεύουσας από την Αλ-Σαμπάμπ, η ίδια η αποστολή Αμισόμ θα κινδύνευε να εξαφανιστεί. Σήμερα αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι εξελίσσεται επιτόπι κατάσταση και βλέπουμε ότι έχουμε τις δυνάμεις της Κένιας οι οποίες υποστηρίζουν τις αρχές του TFG, της μεταβατικής κυβέρνησης, και έχουν προχωρήσει σε στρατιωτικές ε, επιχειρήσεις πολύ σημαντικές στην περιοχή του Γκέντο και του Τζούμπα, έχοντας ως ε, προοπτική να πάρουν την πόλη του Κισμαγιό, που είναι το στρατηγικό λιμάνι, το οποίο εδώ και κάποια χρόνια βρίσκεται στα χέρια της ε, Αλ-Σαμπάμπ. Η προοπτική λοιπόν απελευθέρωση του λιμένα αυτού θα μπορούσε να μετατρέψει πάρα πολύ σημαντικά την, κατάστα την κατάσταση στη Σομαλία. Συνεχίζονται λοιπόν οι προσπάθειες και συνεχίζονται οι συζητήσεις προκειμένου να έχουμε μια νέα αναδιάρθρωση της ε, Αμισόμ. Στην Αντισαμπέμπα την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου έλαβε χώρα μια έκτακτη συνεδρίαση Και ένα από τα συμπεράσματα της συνόδου αυτή ήταν ότι μία από τις καλύτερες εναλλακτικέ που θα είχαμε θα ήταν να συμπεριλάβουμε στην Άμισομ τις δυνάμεις της Κένιας, ενώ η Αιθιοπία θα είχε το δικαίωμα να μπορεί και αυτή να προχωρήσει σε ad hoc επιχειρήσεις υποστήριξης μεταβατικής κυβέρνησης, υποστήριξης της Αμισόμ σε μία εντολή περιορισμένη σε τόπο και χρόνο, χωρίς να αποτελεί αναπόσπαστο και πλήρες τμήμα της ε, αμισόμα. Προσπαθούμε να διευκρινίσουμε λοιπόν καλύτερα αυτή τη νέα προσαρμογή της αμισόμ, προκειμένου να έχουμε μια νέα δυνατότητα επέμβασης. Και προφανώς συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τα Ενωμένα Έθνη, προκειμένου τις επόμενες εβδομάδες ή ακόμα και τις επόμενες μέρες να είμαστε σε θέση να εγκρίνουμε τη νέα αυτή έννοια στρατιωτικής επιχείρησης της Αμισόμ, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος μας είναι να καταφέρουμε να προσαρμόσουμε την εντολή και τις αρμοδιότητες της Αμισόμ στη νέα πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίσουμε επιτόπου. Πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό θα καταφέρουμε να ελοπίσουμε καλύτερα τον οδικό χάρτη όσον αφορά τις, α, τους πολιτικούς στόχους, δηλαδή ένα νέο κοινοβούλιο εκλογές, εκδημοκρατισμός, συμφιλίωση και θα καταφέρουμε επίσης να τονίσουμε και την ανθρωπιστική διάσταση. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες της Σομαλίας που δεν έχουν, που δεν χαίρουν πρόσβαση σε διάφορες ε, ανθρωπιστικές αποστολές, ακριβώς επειδή την πρόσβαση αυτή την εμποδίζουν οι ε, ένοπλες ομάδες της Al-Shabaab. Μπορούμε λοιπόν ότι να πούμε ότι οι νέες αυτές αρμοδιότητες της Αμισόμ θα επιτρέψουν σε πάρα πολλούς Σομαλούς πολίτες να απελευθερωθούν πλέον από τα δεσμά της Al-Shabaab και να έχουν πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Πιστεύουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο η Σομαλία του αύριο θα είναι πιο ειρηνική και θα ενταχθεί στα πλαίσια της συμφιλίωσης και θα δίνονται σε όλους τους Σομαλούς, θα δίνεται σε όλους τους Σομαλούς η δυνατότητα να συμμετέχουν ειρηνικά στην πολιτική ζωή της χώρας. Σχετικά με τη Σομαλία, το θέμα το βασικό της πειρατείας, νομίζω όλοι έχουμε τις ίδιες απόψεις, όποια και αν είναι τα μέσα τα ε, ναυτιλιακά. Ε, μιλάμε για την πειρατεία ε, και τον αντίκτυπό της στη γη. Θα πρέπει να έχουμε διπλή ε, δράση της, της αστυνόμευσης, αλλά και να δούμε και τις, τα αίτια της πειρατείας στην ίδια τη Σομαλία. Ε, και σε στατιωτικό επίπεδο, αν θέλουμε, και να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό στη Σομαλία. Υπάρχουν δύο-τρεις βάσεις πειρατών που θα ε, μπορούσαμε να το κοιτάξουμε από στρατιωτικής άποψης σε αυτή την νέα εντολή που θα υποβάλουμε που ε, περιλαμβάνει και την πειρατεία που αποτελεί μάστιγα και δεν επιτρέπει την ομαλοποίηση της κατάστασης. Άρα η πειρατεία, σε ό,τι μας αφορά, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το χειριστούμε και ε, ε, στο έδαφος της Σομαλίας όχι μόνο στη θάλασσα και πιστεύουμε ότι η Αταλάντα θα πρέπει να έχει επιχειρησιακές σχέσεις κατευθείαν με την Αμισόμ και ε, σε ανατρεπτικό επίπεδο το γεγονός ότι υπάρχει αμισόμ και τα ελικόπτερα της Αταλάντα που ε, υπερίπτανται τις θέσεις της Αμισόν στέλνουν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στην Αρσαμπάπ και τους ε, πείρατες ότι η διεθνής κοινότητα είναι ενωμένη στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και της πειρατείας. Και αυτή η σχέση θα πρέπει να μεταφράζεται από ε, συντονισμένη δράση και ένα εμπάργο ε, της διακίνησης όπλων στην περιοχή αυτή. Με την ίδια ε, δυνατότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή μπορούμε να εφαρμόσουμε ε, το εμπάργο ε, στη διακίνηση όπλων στην περιοχή μέσα από το λιμάνι και το αερολιμένα. Είναι σημαντικό λοιπόν να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή εκεί επί τόπου. Η δικαστική δράση πιστεύουμε ότι πρέπει να οικοδομήσουμε δικαστήρια και φυλακές στην επικράτηση της Σομαλίας. Ε, πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε συμφωνίες με την Κένια, όπως γίνεται μέχρι στιγμής. Όλα αυτά είναι καλά, αλλά δεν αποτελούν λύσεις. Αποτελούν μόνο ad hoc λύσεις, προσωρινές λύσεις. Θα πρέπει να δικαστούν οι Σομαλοί στη Σομαλία με βάση τον Σομαλικό νόμο και να μπορούν να εκτίσουν την ποινή τους στην επικράτεια της Σομαλίας θα πρέπει να ξανακτήσουμε το δικαστικό μηχανισμό στη Σομαλία, ε, δίνοντας στη χώρα τη δυνατότητα να έχουν σοφρονιστικά συστήματα και φυλακές, αλλά είναι μια ευκαιρία να προσπαθούσουμε να δούμε ε, ε, αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν χώροι πέραν του Μογαντήσου, στις, σε άλλες περιοχές υπάρχει δυνατότητα στο κέντρο της Σομαλίας, για παράδειγμα, όπου ε, πάντα υπάρχουν εκεί οι επιδρομές της ε, Al-Shabaab. Υπάρχουν περιοχές, θα μπορούσαν να μας δώσουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε φυλακές και δικαστήρια σε αυτές τις περιοχές που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να λύσουμε τα ε, δικαστικά προβλήματα δικάζοντάς τους ε, στη χώρα τους. Αυτό είναι που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εδώ έγκυται η λύση. Και συνεχώς καλούμε ε, η Αταλάντα να αξιοποιείται έτσι ώστε να ενισχύεται η αποστολή μέσω από άμεσες επιχειρησιακές ε, επαφές. Σε ό,τι αφορά το θέμα της Ομαλίας, ε, η διάσκεψη κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης ζήτησε από ε, το Συμβούλιο Ασφαλείας δύο πράγματα. Ζητήσαμε να έχουμε αποκλεισμό, θαλάσσιο αποκλεισμό είπαν ότι θα πρέπει να υπάρχει συστηματικός έλεγχος και επίσης η ζώνη ενάερου εποπλισμού με ότι δεν μπορούν να υπάρχουν πτήσεις μη εξωστηριοδοτημένων αεροσκαφών που μεταφέρουν, ε, για παράδειγμα, όπλα, χωρίς ε, η κυβέρνηση ή οι άμυσοι να μπορούν να ελέγχουν τα φορτία ή το προσωπικό που μεταφέρεται. Το Συμβούλιο Ασφαλείας όμως δεν έχει ακόμη ε, δώσει σάρκα και ώστα σε αυτά τα αιτήματα. Αλλά μπορώ να σας υποδείξω ότι οι δυνάμεις της Κένιας που βρίσκονται στην Σομαλία αποφάσισαν ότι το αεροδρόμιο Μπάτουα στο οποίο έφτασαν ε, αεροσκάφη γεμάτα οπλισμό ότι θα εφάρμοζαν οι δυνάμεις της Κένιας αυτή την απαγόρευση προσγείωσης οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένου αεροσκάφους από την κυβέρνηση ή την αμισόμη. Υπάρχει συνεχιζόμενη δράση, λοιπόν, με κάποια δημιουργητικότητα. Νομίζω θα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η, η κατάσταση αυτή τη στιγμή έχει κάποια ε, θετικά σημεία. Τέλος, το θέμα του κατακαιρματισμού, όπως γνωρίζετε η Αφρικανική Ένωση και η οργάνωση της ε, στηρίζονται στην ε, αρχή της ανεξαρτησίας και της μη επέμβασης ε, στα σύνορα των άλλων χωρών. Το θέμα του Νοτιού Σουδάν είναι μια εξαίρεση στον κανόνα. Η διάσκεψη αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Αφρικανικής Ένωσης ε, ενέκρινε μία επίσημη απόφαση τον Ιανουάριο του 2010, 11, διορθώνει ο μιλητής, που υπέδειξε ότι για την Αφρική η αρχή της αυτοδιάθεσης δεν πρέπει να εφαρμόζεται παρά μόνο στα εδάφη που βρίσκονται στον κατάλογο των μη αυτόνομων ε, εδαφών της ε, Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δηλαδή στην Αφρική σήμερα υπάρχει μόνο η Δυτική Σαχάρα που έχει το δικαίωμα ε, να επικαλείται την αυτοδιάθεση σύμφωνα με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατοικιαρματισμός είναι το αντίθετο της ολοκλήρωσης. Ενώ εμείς θέλουμε να προωθήσουμε την ολοκλήρωση στην Αφρική. Και κατά τη διαπραγμάτευση της ε, Συμφωνίας για την Ειρήνη, όλα τα μέρη συμφώνησαν για να κάνουν την Ένωση ελκυστική. Όμως βρήκαμε κάποιες δυσκολίες και αναστολές, αλλά όλοι δεσμεύτηκαν να κάνουν την Ένωση ελκυστική. Δυστυχώς αυτό δεν ήταν γιατί ο λαός αποφάσισε να ε, έχει την ανεξαρτησία στο 80% μέσα από το δημοψήφισμα. Μέσα σε 20 χρόνια και για να μειωθούν οι επιδράσεις, οι ενδεχόμενες επιδράσεις τότε αλλά, της, του διαχωρισμού και του κερματισμού ε, ήταν ε, το γεγονός ότι θα δημιουργούνταν κράτη που θα ε, συμπίωναν ειρηνικά το ένα δίπλα στο άλλο, δημιουργώντας ε, συνέργειες και συνεργασίες ανάμεσα στα δύο κράτη. Και αυτό αντιμετωπίζουμε σήμερα. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα που εκκρεμούν, αλλά πρέπει, ε, χρειάζεται πολύ κουράγιο και δημιουργικότητα και φαντασία. Η Αφρική και η διεθνής κοινότητα ε, πρέπει να τοποθετηθούν σαφώς αυτό το πελαίσιο όταν ε, πρόκειται για τα προβλήματα της Σομαλίας. Θα πρέπει να ε, εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι σχεδόν σε όλες τις αφρικανικές χώρες όπου υπάρχουν προβλήματα η πρόκληση είναι πώς να εναρμονίσουμε την ενότητα και την διαφορετικότητα και να πετύχουμε την ε, δημοκρατικοποίηση, την πλουραλιστική, που θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε την ενότητα, διατηρώντας τη διαφορετικότητα. Οι συνταγματικές δομές που ξέρουμε, οι ομοσπονδίες θα μπορούσαν επίσης να ε, λάβουν υπόψη αυτά τα θέματα, ιδιαίτερα στη Σομαλία, όπου έχουν επιτευχθεί κάποια επίπεδα ανάπτυξης, και μπορεί να μην έχουν τη σταθερότητα που έχουν άλλες περιφέρειες, αλλά και εκεί θα μπορούσαν να ενευρεθούν λύσεις. Και είναι γι' αυτό που η δράση της εκπόνησης του στάγματος της Σομαλίας με τη συμμετοχή όλων ε, δυστυχώς ε, δεν ήταν όλοι παρόντες το Σεπτέμβριο ε, ελπίζουμε ότι θα είναι στην επόμενη φορά και όλες αυτές οι περιφέρειες θα συμμετέχουν έτσι ώστε ε, το συνταγματικό μέσο που θα δημιουργηθεί με βάση την ηθαγένεια και την ισότητα των υπηκών θα διευθετήσει αυτό το μέσο όπου όλοι θα αισθάνονται άνετα στο κράτος της Ομαλίας και θα δώσει σε όλους τους πολίτες ένα καλύτερο μέλλον από αυτό το οποίο έχει ζήσει μέχρι στιγμής ε, η χώρα. Τέλος, νομίζω ότι θα πρέπει να πω και κάτι για το Σαχέλ και για την Αραβική Άνοιξη. Πρώτα απ' όλα για το Σαχέλ. Εμείς στην Αφρική Ένωση χαιρόμαστε που τα κράτη της περιφέρειας ε, οργανώθηκαν και ανάπτυξαν ένα σαφές όραμα και προσανατολισμένο προς την κοινή δράση με βάση μια κοινή αντίληψη των κινδύνων και επίση χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει το στρατηγικό πλαίσιο για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στην περιοχή του Σαχέλ. Ένα έγιναν αρκετές επαφές ε, και στα πλαίσια της ομάδας εργασίας ε, από το Παγκόσμιο Φόρουμ κατά της τρομοκρατίας και πιστεύουμε ότι σήμερα περισσότερο ότι ποτέ στο, παρελθόν έχουν τεθεί τα προβλήματα του Σαχέλ και όταν τοποθετούνται σωστά τα προβλήματα μιας ε, περιοχής, τότε είμαστε πιο κοντά στην αντίληψη των ε, θεραπείων στα προβλήματα. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των ε, μέσων που έχουμε την καταπολέμηση της τρομοκρατίας έχουμε συνεισφέρει σε αυτό το τομέα. Εκεί πάλι πρόκειται για ενισχυμένη συνεργασία, όπως και στην άλλη πλευρά της ε, Αφρικής, ε, όπως κατά πολέμηση του LRA, του Αντιστασιακού Στρατού του Κυρίου. Και αυτό αποδεικνύει το έργο της Αφρικής με τα διάφορα περιφερειακά όργανα και τα εθνικά όργανα για την καταπολέμηση των επιδράσεων αλλά και των βαθέων αιτίων, βαθιών αιτίων ε, των καταστάσεων αυτών. Πράγματι, η Λιβύη το τελευταίο μήνα ε, αποτελεί μια ε, ένα ένα, μια αποθήκη πυρομαχικών, αν θέλετε, και έχουν ανεβρεθεί ε, πολλά ε, όπλα σε αυτή την περιοχή ε, με κίνδυνο σε όλη την περιοχή του Σαχέλ και διακίνηση όπλων σε όλη την περιοχή. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε με τις νέες αρχές της Λιβύης με όλες τις γειτονικές χώρες και τη διεθνή κοινότητα και τους διεθνείς οργανισμούς που εξειδικεύονται στον έλεγχο της διακινήσης όπλων για να οργανώσουμε συνεργασίες με στόχο την συλλογή αυτών των όπλων και να παρεμποδίσουμε ε, την ε, περαιτέρω αστάθεια στην περιοχή. Είμαστε σε επαφή με τα τον ΟΗΕ, τον Αραβικό Σύνδεσμο και τις αρχές της Λιβύης και τις διάφορες γειτονικές χώρες ε, στα ζητήματα αυτά που αποτελούν κλειδί για τη σταθερότητα του χώρου της Μεσογείου αλλά και του χώρου της του, περιοχής του Σαχέλ και της υποσαχάριας Αφρικής. Αραβική Άνοιξη θα είμαι πολύ σύντομος γιατί πρώτα απ' όλα είναι επίμαχο κατά πόσο α, αυτός ο όρος είναι σωστός. Νομίζω είναι πολύ πιο περίπλοκο το φαινόμενο αυτό που παρατηρείτε. Τώρα, κατά πόσο θα έχει επιπτώσεις, ίσως όχι στους βασικούς κανόνες της ε, στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρική, αλλά στις ανησυχίες, στον τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας, ε, γιατί οι πρόοδοι της δημοκρατίας θα έπρεπε πάντα να αποτελούν θετικές βάσεις για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των στόχων, των κοινών μας στόχων. Για τον Νότιο Σουδάν, με μια λέξη, το Νότιο Σουδάν έχει τις προκλήσεις οποιοδήποτε νέου δημοκρατικού κράτους. Μεγάλες προκλήσεις, όπως είπα, ε, για να μπορέσει να διευθετήσει ορισμένα ε, θέματα που εκκρεμούν. Ε, δυστυχώς γίνεται ένα βήμα μπρος και δύο πίσω, όπως η κατάσταση του πετρελαίου που πρέπει να λυθεί. Αυτή τη στιγμή έχει μόνο μία διέξοδο προς το βόρειο Σουδάν, θα πρέπει να βρει λύσεις, βέλτιστες λύσεις για να μπορέσουν αυτά τα δύο κράτη να βρουν συνεργασία με κοινά συμφέροντα. Υπάρχουν και άλλοι τομείς στον τομέα της ασφάλειας, στον τομέα της ε, πολιτικής ζωής, ε, χωρίς ε, να υποστηρίζονται οι στρατιωτικές ε, δυνάμεις της μιας και της άλλης ε, χώρας. Ε, δημοκρατική Δημοκρατία του Κόγκο είχαμε χθες εκλογές, συνεχίζουν να ψηφίζουν και σήμερα. Έχουμε ίσως αποφύγει το χείριστο. Το ελπίζουμε σήμερα θα είναι η δοκιμασία, δηλαδή η καταμέτρηση των ψήφων και η αποδοχή των αποτελεσμάτων όταν ανακοινωθούν αυτά. Ε, είμαστε επιτόπου και εμείς έχουμε παρατηρητές εκεί. Έχουμε μεταβεί για να τον τριασμό της κατάστασης και την αποδοχή ε, των αποτελεσμάτων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Ζαμπίν, ήταν εκεί και είναι σαφές ότι η επιτυχία της διαδικασίας, της δημοκρατικής διαδικασίας ε, στο Κόγκο θα έχει αντίκτυπο και στις γειτονικές χώρες ε, και στην Ήπειρο της Αφρικής γενικά, ακόμη και αν η διαδικασία έχει κάποιες αδυναμίες λόγω της υποανάπτυξης, αλλά αυτή είναι η τάση που πρέπει να ακολουθείτε και ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα, όποια και αν είναι, θα γίνουν αποδεκτά από όλα τα κόμματα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη, κύριε Γενική Διευθυντή, ενδεχομένως σύντομα εσείς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πέντε σύντομε παρατηρήσεις. Καταρχάς, το ζήτημα του κυρίου Γκολτιέρη για τους πόρους. Ήδη χρησιμοποιούμε τον φορέα σταθερότητα ε, και μέσω αυτού όταν θέλουμε να επέμβουμε άμεσα με υποστηρικτικά μέτρα χρησιμοποιούμε αυτό το φορέα ή άλλα ταμεία ή το IFS. Επίσης, ε, ε, το η υποστήριξη από πλευράς EDF πρέπει να είναι ευέλικτη, διότι μόνο αν εξασφαλιστεί η σταθερότητα μπορούμε να εξασφαλίσουμε και την ανάπτυξη. Ε, άρα λοιπόν μέσω του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου χρησιμοποιούμε πόρους και από εκεί. Για τη Σομαλία είναι σωστό ότι υπάρχει ο κίνδυνος εξωτερικής παρέμβασης, ότι θα δώσει τη δυνατότητα στην Al-Shabaab να δρέψει εθνικιστικές δάφνες ε, εναντίον των εξωτερικών επεμβάσεων δηλαδή να χρησιμοποιήσει εθνικιστικά συνθήματα και προπαγάνδα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα προς την Αιθιοπία, για το πώς θα μπορέσει να προσφέρει υποστήριξη στην ε, TFG, για να μην ε, οξύνουμε περισσότερο τους κινδύνους. Είναι σαφές ότι η Al-Shabaab παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη οργάνωση. Έχει, μόλις κατάφερε να διώξει τη UNICEF και άλλους φορείς βοήθειας ε, προς το πληθυσμό, τους πέταξε έξω από τις περιοχές της, ε, από τις περιοχές που ελέγχει και και δεν ενδιαφέρεται ουδόλως για την ευημερία ή τέλο πάντων τη βοήθεια προς τον άμαχο πληθυσμό. Είναι λοιπόν λίαν επίγον να βρεθεί μία ε, πολιτική λύση για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον λιμοκτονούντα πλησισμό αυτής της περιοχής. Όσον αφορά τώρα την πειρατεία, πολλά γίνονται. Πολλά γίνονται. Ε, αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε τις ε, διαβουλεύσεις μας ε, και στο, με την Μαυριτανία και με την Τανζανία για τη μεταφορά των συλληφθέντων έτσι να μπορούν οι πειρατές να, δικαστούν. Να τους δικάσουμε σε δικαστήρια. Επίσης λειτουργούμε ε, εν πλήρη αρμονία με τις άλλες δυνάμεις ε, εδάφους, παρόλο που η πειρατεία βεβαίως είναι στη θάλασσα και όχι στην ξηρά. Όμως πρέπει να διατηρούμε και ε, επιχειρήσεις στη θάλασσα αλλά και στην ξηρά. Έχω έχουν γίνει ε, πολλές, έχουμε σημειώσει επιτυχία στην αποφυγή επιθέσεων και κατάληψη σκαφών και η κατάσταση έχει βελτιωθεί από τα προηγούμενα δύο χρόνια. Υπάρχει μία πρόοδος ε, σχετική, δεν είναι μόνιμη αυτή η λύση, αλλά οι Υπουργοί Εξωτερικών έχουν συμφωνήσει να ορίσουν έναν ε, ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κέρας της Αφρικής για να μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα μέσω της υπηρεσία αυτής και του, του ατόμου αυτού, της θέσης αυτής, να επιληθούν καλύτερα τα προβλήματα. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει να βρούμε μια ισορροπη, ισορροπημένη πολιτική λύση για όλη την περιοχή και στην Σομαλία, όπως είπε και ο πρέσβης ε, κύριος ε, Λαμάμρα. Ε, πρέπει να βρούμε μια δομή κατάλληλη που να καλύπτει όλες τις ανάγκες. Και κάθε διαβούλευση που γίνεται προς αυτό το στόχο την υποστηρίζουμε. Επίσης, πιστεύω πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα για το Σουδάν ε, να υπάρξουν δύο κράτη. Όμως και το Βόρειο και το Νότιο έχουν τεράστια προβλήματα και θα πρέπει και τα δύο κράτη αυτά να δεσμευτούν ως προς την εξέβρεση ειρηνικής λύσης. Και οι δύο πλευρές πρέπει να έχουν καταλάβει μέχρι τώρα ότι ο πόλεμος και η συνεχή σύραξη δεν είναι λύση και θα πρέπει στην Άντιγε και σε όλες τις περιοχές αυτές αυτές ε, να λύσουν τα συνοριακά προβλήματα. Όσον αφορά τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό τώρα και πάλι η προσέγγιση μας είναι ε, σύμφωνη με αυτή που εξέθεσε ο κύριος Πρέσβης. Τα γεγονότα τα στη Βάρη Αφρική, αν θέλετε ονομάστε την Αφρικανική Άνοιξη, έδειξαν ότι δεν υπάρχει, δεν, δεν είναι φρόνιμο να παραποιήσει κανείς τα εκλογικά αποτελέσματα, να νοθεύσει τις εκλογές, διότι δεν, οδηγεί σε, δεν έχει κανένα θετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό οι νοθευμένες εκλογές δεν επιτυχάνουν τίποτα. Δεύτερον, δεν ε, είναι δυνατόν να στα, κρατηθεί στην εξουσία SAE όταν συνεχίζεις να σφάζεις και να σκοτώνεις τους δικούς σου πολίτες. Γι' αυτό οι χώρες αυτές που οργανώνουν τέλος πάντων εκλογές στη Βόρεια Αφρική σήμερα, αύριο, μεσάβριο, βασμιαία λοιπόν θα επιβληθεί ένα εκλογικό σύστημα μετά από τα παθήματα, τα παθήματα μαθήματα. Τρίτον, ε, απογοητεύτηκα ε, πολύ προσωπικά από το μποϊκοτάζ των εκλογών, του, του δεύτερου γύρου των εκλογών στη, Λιβερία. Δεν είναι σωστή διαδικασία αυτή. Δεν είναι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε στη Λιβερία. Ελεύθερες και δίκαιες εκλογές είναι ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε. Μία κατεύθυνση υπάρχει, μόνο μονόδρομος και δεν υπάρχει ε, δεν είναι δυνατόν να μην γίνει αποδεκτό το αποτέλεσμα των εκλογών, διότι ε, σε περιφερειακό επίπεδο και οι γειτονικέ χώρε δεν θα δεχθούν αυτή την κατάσταση ανατροπή των εκλογών. Επίση για την ε, Σαχέλ δεν έχω να πω πολλά περισσότερα, διότι τα εξέθεσε πάρα πολύ καλά εκπρόσωπο και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων που ήταν πολύ χρήσιμη για μένα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Διευθυντή, κύριε Πρέσβη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανοιχτή, ανοιχτή αυτή συζήτηση που είχαμε μαζί σας. Μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να καταλάβουμε καλύτερα την εργασίες της Επιτροπής σας και τη συνεργασία που έχετε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα δύο λεπτών προτού προχωρήσουμε στο επόμενο τμήμα της μας που έχει να κάνει με το Σαχέλ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Καθίστε σας παρακαλώ πολύ. Καθίστε σας παρακαλώ όλοι και οι εξωτερικοί παρατηρητές. Το δεύτερο αυτό τμήμα της συνεδρίασής μας έχει να κάνει με την Αφρική, με μια περιφέρεια με την οποία ασχολούμαστε πολύ συχνά στην υποεπιτροπή μας, την περιφέρεια του Σαχέλ, που τις τελευταίες μέρες είχε τραγικές εξελίξεις για τους Ευρωπαίους πολίτες Τέσσερις Ευρωπαίοι πολίτες ε, έπεσαν θύμα απαγωγής, ένα σκοτώθηκε, στο Μαρί συγκεκριμένα. Βλέπουμε λοιπόν κάθε μέρα ποιος είναι ο πραγματικός αυτός χαρακτήρας της τρομοκρατικής απειλής ε, στην περιοχή αυτή, τρομοκρατική απειλή για την οποία θέτουμε πάρα πολλά ερωτήματα, ιδίως μετά τις εξελίξεις στη Λιβύη, και ιδίως μετά τα όσα λέγονται για τις έντονες μετακινήσεις ε, όπλων αλλά και στρατιωτών μεταξύ των συνόρων, στα νότια δηλαδή της ε, Λιβύης και με, στην περιοχή του Σαχέλ. Στις 29 Μαρτίου το Συμβούλιο κατέληξε σε μια στρατηγική για το Σαχέλ. Περιλαμβάνονται τέσσερις βασικοί άξονες. Η ασφάλεια και η ανάπτυξη είναι έννοιες ε, που συνδέονται και είναι απαραίτητε για το Σαχέλ. Εμείς άλλωστε στην Επιτροπή μας πάντα συνδέουμε την έννοια της ασφάλειας με την έννοια της ε, ανάπτυξης και θα έχουμε και τη δυνατότητα να μιλήσουμε περισσότερο με τον κύριο Κερκόφ και τον κύριο Λοπές Μπλάνκο. Έχουμε επίσης ε, το ζήτημα της περιφερειακής συνεργασίας. Έχουμε καταφέρει να σημειώσουμε πρόοδο. Πολλές φορές η πρόοδος αυτή είναι απλώς διακοσμητική, άλλες φορές όμως καταδεικνύει την πραγματική βούληση των κρατών της περιοχής να συνδεθούν περισσότερο, να συνεργαστούν περισσότερο. Πρέπει επίσης να ενδυναμώσουμε, να ενισχύσουμε τις κρατικές ικανότητες, το κρατικό δυναμικό το οποίο υπάρχει όσον αφορά την στρατιωτική και αστυνομική δύναμη και ένας τέταρτος και τελευταίος άξονας, ο ρόλος που θα μπορέσει να δραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να υποστηρίξει τις εξελίξεις αυτές, συνδέοντας ακόμα περισσότερο την έννοια της ασφάλειας με την έννοια της ανάπτυξης. Έχουμε μαζί μας τον Ζιλ Τεγιακόφ, ο οποίος είναι ο συντονιστής της αντι... αντιτρομοκρατικής δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γνωρίζουμε καλά και τον ευχαριστούμε που έχει έρθει, τον ευχαριστούμε μάλλον που έρχεται πολύ συχνά και μας ενημερώνει για την εξέλιξη στην περιφέρεια αυτή και μπορούμε χάρη στη δική του παρέμβαση να γνωρίζουμε πώς βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις εξελίξεις ε, στην ε, περιοχή αυτή και έχουμε και τον κύριο Φιλιμπέρτο Τσεριάνη Σεμπρεγκόντι, ο οποίος αντικαθιστά τον Μανουέλ Λόπες Μπλάνκο και εκπροσωπεί εδώ πέρα την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Μπλάνκο δεν κατάφεραν σήμερα μαζί μα. Πολύ σύντομα θα εκπροσωπήσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τανζανία, αλλά σε έχουμε καλέσει εδώ πέρα κυρίω για τι γνώσει που έχετε για την περιοχή του Σαχέλ. Ευθύ αμέσω να δώσω το λόγο στον κύριο Ντεκερκόφ και στη συνέχεια στον κύριο Τσεριάννη Ζεμπραγκόνη. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που με καλείτε συχνά. Όντω ε, βρίσκω και εγώ ότι η ανταλλαγή απόψεων που έχουμε είναι πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ πολύτιμη καταφέρνουμε κατά αυτόν τον τρόπο να σας λέμε με τον πλέον διαφανή τρόπο τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει και να αξιολογήσει τον κίνδυνο. Όσον αφορά τη στρατηγική Σαχέλ, θα ήθελα να αφαιρθώ σε αυτήν και συνέχεια να αφαιρθώ στις νέες εξελίξεις, στις οποίες αναφερθήκατε και εσείς, Πρόεδρε, και τέλος να σας πω πώς θα λάβει υπόψη της Ευρωπαϊκή Ένωση τις νέες αυτές εξελίξεις. Τον Μάρτιο οι ε, Υπουργοί Εξωτερικών κατέληξαν σε μια στρατηγική για το Σαχέλ, η οποία, και το λέω αυτό συνεχώς, Ακούγεται κοινότοπο, αλλά πραγματικά η στρατηγική αυτή είναι καινοτόμα. Πρώτη φορά προσπαθούμε στα πλαίσια τη ίδια στρατηγική να συνδυάσουμε ασφάλεια και ανάπτυξη. Δεν είναι αυτονόητο το ζήτημα αυτό και πολύ πιο δύσκολο όταν εφαρμόζεται επιτόπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω να συνδυαστεί η ασφάλεια με την ανάπτυξη και αν καταφέρουμε στην πράξη να ελοποιήσουμε τη διασύνδεση του Σαχέλ, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πολύ θετικό προηγούμενο το οποίο θα μπορεί να εφαρμοστεί και στι άλλε περιφέρειες Αφρική, αλλά και σε όλε τι περιοχέ του κόσμου. Ακούσαμε τον πρέσβη Λαμαμάρα πριν από λίγο και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι να εφαρμοστεί αυτό και στις άλλες περιοχές. Αναφερθήκατε στις, στους τέσσερις βασικούς άξονες της στρατηγικής. Στο Αλγέρι, σε αρχές Σεπτεμβρίου, σε μια συνάντηση, είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πραγματική ηγετική θέση στην περιφέρεια της ε, Αφρικής χρειάστηκε να ταφανίσει πάρα πολύ χρόνο, αλλά έχουμε πλέον μια, ένα σαφή ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αφρικανική Ήπειρο. Πολλά μέλη του ΚΟΠΣ, της Πολιτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης, και της εξωτερικής πολιτικής πραγματικά καταφέρνουμε να έχουμε ένα συντονισμό όλων των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε πρόκειται για δράση κρατών μελών, είτε πρόκειται για δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε πρόκειται για τα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. 400 εκατομμύρια δίνουμε στον Ήγυρα, το Μαλί, τη Η στρατηγική λοιπόν του Σαχέλ ήδη έχει οδηγήσει σε αυτή την κινητοποίηση των 150 εκατομμυρίων φρέσκων πόρων, θα έλεγα, που ε, βρίσκονται σε φάση δέσμευση. Το Μάρτιο εγκρίθηκε η στρατηγική του Σαχέλ, αλλά εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο το οποίο υπήρχε ήδη στο παρελθόν. Προσπαθούμε απλώ να γενιάσουμε τώρα κάποια νέα προγράμματα. Ο συνάδελφό μου θα σα δώσει περισσότερε πληροφορίε. Εγώ ασχολούμαι περισσότερο με το ζήτημα τη ανάπτυξη. Συνάψαμε επίσης διάφορες συμβάσεις και συμφωνίες στον Νίγηρα υποστήριξη για παράδειγμα για το κράτος δικαίου και για το δικαστικό σύστημα, η υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών για τη βελτίωση του διαλόγου ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες κοινωνίας των πολιτών, μια έκτακτη χρηματοδότηση 12 εκατομμύρων ευρώ, δεν θα προχωρήσω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι η δράση μας είναι τόσο σημαντική όσο για την ανάπτυξη, όσο όμως και για την ασφάλεια. Έχουμε σε μια πρώτη φάση 835 εκατομμύρια ευρώ και 6,7 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν σε μια δεύτερη βάση για το Μαλί, τη Μαυριτανία και για το Νίγηρα τώρα. Προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία και για τη χώρα αυτή. Καθυστερήσαμε λίγο γιατί η χώρα βρίσκεται σε φάση εκδημοκρατισμού. Έχουμε μία παραδοσιακή προσέγγιση όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας, καλύτερη συλλογή και μεταχείριση των δεδομένων από πληροφοριακής άποψης, καλύτερη βελτίωση της ποινική αλυσίδας, καλύτερη συνεργασία των αστυνομικών δυνάμεων, των δικαστικών δυνάμεων και καλύτερη διαχείριση των κρίσεων από τις αρμόδιες ομάδες στη χώρα. Αυτό το οποίο είναι πιο σημαντικό πέρα από την παραδοσιακή αυτή προσέγγιση είναι να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα κολέγιο ασφάλειας για την καλύτερη ενημέρωση των διαφόρων ε, ομάδων που δρούν για την ασφάλεια στην περιοχή του Σαχέλ, αλλά και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο επίπεδο εμπιστοσύνης. Ξέρετε ότι ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την ενημέρωση, την κατάρτιση και αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει σε μια καλύτερη συνεργασία. Το κολέγιο αυτό, η ακαδημία αυτή, είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά αρχίζει και υλοποιείται, βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή, θα μπορούσε να ενδυναμωθεί από άλλες αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποστολές εξωτερικής δράσης και ουσιαστικά θα κινητοποιήσει διάφορους φορείς υπεύθυνους για την ασφάλεια στην περιοχή και συνδέεται με το ΣΕΜΟΠ και το ε ΕΦΕΛ, τις πρωτοβουλίες δηλαδή ασφάλεια στην περιοχή που δημιουργήθηκαν στην Αλγερία. Ποιες είναι τώρα οι τελευταίες εξελίξεις. Τρεις σημαντικές έχουμε. Πρώτον, οι συνέπειες των όσων συνέβησαν στη Λιβύη, η ε, ανάπτυξη δυστυχώς περαιτέρω εξέλιξη της ΑΚΜΗ, καθώς επίσης ε, και η ε, εξελίξεις που έχουμε στον αραβικό κόσμο, στι οποίε αναφερθήκαμε πριν από λίγο. Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, σαφώ υπάρχει μετά την ε, αλλαγή του καθεστώτος στην ε, Λιβύη μια διάδοση διαφόρων όπλων, διαφόρων ειδών οπλισμού, αφορητού οπλισμού, ελαφρού οπλισμού, εκρηκτικού, ε, εκρηκτικών μηχανισμών. Στις 12 Ιουνίου καταφέραμε να σταματήσουμε στον Ήγυρα 672 κιλά πυρομαχικών μέσα σε ένα φορτηγό. Δεν έχουμε ακόμα μια ξεκάθαρη ακριβή εικόνα της κατάστασης. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ καμένα από τη Λιβύη όσον αφορά τα πυρομαχικά, όσον αφορά τα απλοστάσια, όσον αφορά τα όπλα τα οποία διακινούνται από τη χώρα αυτή προς άλλες χώρες. Έχουμε βέβαια διάφορες πληροφορίες οι οποίες ε, καταδεικνύουν ότι προφανώς τα φαινόμενα αυτά δεν περιορίζονται στην ε, Λιβύη. Προφανώς θα πρέπει να αφοπλιστούν οι παραστρατιωτικές ε, οργανώσεις αλλά θα πρέπει να συλλεχθούν και τα όπλα αυτά τα οποία έχουν κινηθεί από την Λιβύη προς ε, διάφορες χώρες ε, του Σαχέλ που χρησιμοποιούνται ουσιαστικά στην δευτερογενή αγορά και πολλές φορές καταλήγουν ακόμα και στα χέρια της ΑΚΜΗ, της Αλκάιντα δηλαδή στον Ισλαμικό, στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ. Επίσης ε, Έχουμε διάφορους μισθοφόρους οι οποίοι μετά τις δράσεις τους στη Λιβύη επέστρεψαν στις χώρες τους. Πολλές χώρες ε, χρειάστηκε να επαναπροφήσουν 200 με 250 χιλιάδες τέτοιους άνεργους. Αυτό αποτελεί μια πάρα πολύ σημαντική πρόκληση που μπορεί να οδηγήσει στην αποσταθεροποίηση περισσότερο της περιοχής και ιδίως του Νίγηρα. Να αναφερθώ επίσης και στην ΑΚΜΗ, στην Αλκάιντα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ. Έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια. Τέσσερις ή πέντε εξελίξεις έχουμε. Έχουμε μια γενικότερη τάση αφρικανοποίησης της ΑΚΜΗ στην Κεντρική Αφρική. Ξεκίνησε ουσιαστικά από την Αλγερία. Είχε συναντήσει πολλές δυσκολίες στην αρχή κατάφερε όμως να ανασυνταχθεί και βλέπουμε ότι δεν έχει ακόμα μία απόλυτη ανεξαρτησία, αλλά βλέπουμε ότι καταφέρνει και κερδίζει όλο και μεγαλύτερη αυτονομία σε σχέση με τις αλγερινές ρίζες της και έχει όλο και μια μεγαλύτερη διασύνδεση με την Αλκάιντα του Πακιστάν. Μια γενικότερη τάση, ιδιαίτερα ενισχυτική και αυτή, είναι ότι στι ζώνε όπου έχει εξαφανιστεί ο κρατικό μηχανισμό και όπου οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πολλέ δυσκολίε, η ΑΚΜΗ τελικά έχει αναλάβει μια δράση τύπου Χεσμπολά. Δηλαδή, παρέχει διάφορε κοινωνικέ υπηρεσίε, αγοράζουν διάφορα τρόφιμα τα οποία στη συνέχεια πουλάνε δύο-τρεις φορές περισσότερο στους ε, κατοίκους προχωρούμε σε διάφορες δραστηριότητες επίβλεψης, επιτήρησης κτλ. Τρίτον, βλέπουμε ότι η ακμή δεν γίνεται ακόμα μία καθαρά εγκληματική οργάνωση, διατηρεί ακόμα κάποια στοιχεία ιδεολογίας, αλλά συμμετέχει σε διάφορα εγκληματικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα η διακίνηση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαίνης. Έχουν καταφέρει να στρατολογήσει περισσότερους μαχητές, έχουν καταφέρει να επεκταθεί γεωγραφικά σε διάφορες περιοχές και ανησυχούμε επίσης γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πλέον και διάφορες διασυνδέσεις με αραβικές ομάδες όπως για παράδειγμα η Άλλα Σαμπάμπα. βλέπουμε ότι η συνεργασία τους με ορισμένες τρομοκρατικές ομάδες της Αφρικής είναι ιδιαίτερα διαρθρωμένη. Θα αναφερθώ περισσότερο στην ομάδα αυτή, η οποία βρίσκεται στον Βόρειο Νίγηρα. Ήμουνα στην χώρα αυτή μαζί με τον κύριο Μπλανκό την προηγούμενη εβδομάδα και θα σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν, η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε στον Βόρειο Νίγηρα, στην Βόρεια Νιγηρία, με συγχωρείτε, στην περιοχή Μπορνό και Γιομπέ. Πρόκειται για Ταλιμπάν της Νιγηρίας τελικά που θέλουν να δημιουργήσουν ένα καθαρό Ισλάμ, το οποίο θα εφαρμόζει πολύ αυστηρά τον Ισλαμικό νόμο της Σαριά. Θα έλεγα ότι έχουν μια τοπική ατζέντα, κάποιες τοπικές προτεραιότητες. Υπάρχουν ορισμένοι που έχουν χρησιμοποιηθεί από διάφορους ε, τοπικούς πολιτικούς προκειμένου να καταφέρουν να προωθήσουν τη δική τους πολιτική ατζέντα. Ε, ασχολούνται με διάφορες συνήθεις εγκληματικές δραστηριότητες. Ε, έχει καταφέρει να δημιουργηθεί η ομάδα αυτή στα πλαίσια μιας απόλυτης φτώχειας, ένδυας, καταστροφής του περιβάλλοντος, ε, με έντονες ε, σχέσεις αντιπαράθεσης με διάφορες όμορες χώρες όπως ο Νίγηρας ή το Τσάντ. Είπαμε ότι απουσιάζει πάρα πολύ ο κρατικός μηχανισμός, όπως γενικότερα βλέπουμε στην περιοχή του Σαχέλ και τους τελευταίους μήνες η ομάδα αυτή έχει καταφέρει να αυξήσει τη δύναμή της μέσω των διαφόρων επιχειρήσεών της, των διαφόρων επιθέσεων αυτοκτονίας που δεν είχαμε στο παρελθόν στην περιοχή αυτή. Ουσιαστικά μιμούνται τον τρόπο λειτουργίας της Αλκάιντα και έχουν κατα... μάλλον καταρτίστηκαν ορισμένοι στα πλαίσια και άρχισαν να επικεντρώνονται σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς. Είχαμε για παράδειγμα μια δολοφονική επίθεση στην Αμπουτζά στον κτίριο των Εθνών με 26 νεκρούς καθώς επίσης και μια επίθεση στο Γενικό Επιτελείο των Αστυνομικών Δυνάμεων στο, στην Ιγυρία. Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, αυξάνουν γενικότερα την δύναμή τους και την παρουσία τους και πρέπει λοιπόν να επικαιροποιήσουμε την στρατηγική του Σαχέλ που εγκρίθηκε το Μάρτιο, που αναφερόταν στρατηγική στο φαινόμενο αυτό, αλλά βλέπουμε το φαινόμενο αυτό έχει από τότε εντατικοποιηθεί. Να αναφερθώ και στις συνέπειες της κρίσης στη Λιβύη όσον αφορά τη διάδοση των όπλων Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τους Αμερικανούς μας συναδέλφους, οι οποίοι ε, πολύ γρήγορα μετά την απελευθέρωση της Τρίπολης απέστειλαν εμπειρογνώμονες επιτόπου, εξειδικευμένες ομάδες προκειμένου να εντοπιστούν τα πυρομαχικά, οι πύραυλοι, να καταφέρουμε να προστατεύσουμε περισσότερο συγκεκριμένα μέρη της ε, Λιβύης. Ε, συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τις με τα Ηνωμένα Έθνη στα πλαίσια της ανοικοδόμησης της Λιβύης. Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται τα εξωτερικά σύνορα, υποστηρίζει την κοινωνία των πολιτών και τα Ηνωμένα Έθνη ασχολούνται περισσότερο με τις διαδικασίες ε, ε, ε, ολοκλήρωσης. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα καταφέρουμε να αποστείλουμε εμπειρογνώμονες και η κυρία Άστον ασχολείται εκ του σύνεγγης με το ζήτημα αυτό, είχε πάει μάλιστα και στην Λιβύη πρόσφατα. Βλέπετε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει πραγματικά να υποστηρίξει την ανοικοδόμηση τη χώρα. Όσον αφορά τώρα το Σαχέλ, και ο συνάδελφό μου θα σα πει περισσότερα πράγματα. Προσπαθούμε βραχυπρόθεσμα να ενισχύσουμε το μέσο σταθεροποίησης με την έγκριση ενός πακέτου το οποίο θα κινητοποιηθεί πολύ γρήγορα τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου, 9 εκατομμύρια περίπου θα δοθούν στην περιοχή, προκειμένου να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τις χώρες της περιοχής αυτής να υλοποιήσουν το σχέδιο ασφάλειας και ανάπτυξης για το βόρειο ε, Νίγηρα και προκειμένου να ληφθούν κάποιες βραχυπρόθεσμες άμεσες αποφάσεις για την ενσωμάτωση των μαχόμενων. Θέλουμε, για παράδειγμα, να τους εντάξουμε περισσότερο σε κάποιες τοπικές αστυνομικές δυνάμεις, να ασχοληθούν με την αρκαλίευση, να υποστηρίξουν κάποιες οικονομικές δυνατό, κάποιες, κάποιους οικονομικούς τομείς που έχουν ανάγκη από χέρια. Αυτές είναι οι επιπτώσεις λοιπόν της ε, κατάστασης στη Λιβύη. Πιο συγκεκριμένα για το Σαχέλ, τους τελευταίους μήνες γίνανε πολλές ε, διεθνείς ε, συνεδριάσεις που μας επέτρεψαν και να εξηγήσουμε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και να δημιουργήσουμε συμμαχίες. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μια πρωτοβουλία ιδιαίτερα χρήσιμη του πρώην Υπουργού Εσωτερικών Ουμπαλκαμπά της Ισπανίας, όπου συνεδριάζουν οι έξι υπουργοί εσωτερικών των πιο πυκνοκατοικημένων κρατών στη Μαδρίτη, προκειμένου να υπάρχει μια πιο έντονη συνεργασία μεταξύ τους. Υπάρχει λοιπόν συνεργασία ανάμεσα στα Υπουργεία Εξωτερικών, τα Υπουργεία Δικαιοσύνη και αν πραγματικά θέλουμε να στείλουμε εμπειρογνώμονε πρέπει πρώτα να εντοπίσουμε του καλού αυτού εμπειρογνώμονε στην Ευρώπη, πρώτα του στείλουμε στην Αφρική. Είχαμε έπειτα και τη συνδιάσκεψη τη Αλγερία που έγινε με πρωτοβουλία τη Αλγερία, του Μαλή, του Νίγηρα και τη Μαυρετανία αρχέ Σεπτεμβρίου του 2011, εγώ συμμετείχα μαζί με τον συναδελφό μου κύριο Μπλάνκο και ήταν η πρώτη σημαντική διεθνής συνδιάσκεψη κρατών της περιοχής αυτής που ανοίγονταν ουσιαστικά για πρώτη φορά προς τη διεθνή κοινότητα. Και θέλαμε να δούμε από κοινού τι μπορούσαμε να κάνουμε για την περιοχή. Το μήνυμα το οποίο στάλει ήταν πολύ θετικό, γιατί εδώ και δύο-τρία χρόνια το κλίμα δεν ήταν ιδιαίτερα ευέλικτο και ανοιχτό. Η Αλγερία, για παράδειγμα, ήταν πάρα πολύ διστακτική απέντη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ήθελε να συμμετέχει άμεσα ή έμεσα στο, στην πολιτική του Σαχέλ. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τέσσερις χώρες να συνεργάζονται, τέσσερις κυβερνήσεις να επιθυμούν από κοινού να επιλύσουν κάποια προβλήματα. Και πάλι συμπενθυμίζω ότι πριν από δύο χρόνια υπήρχε ένας πολύ υψηλός βαθμός δυσπιστίας ανάμεσα στις τέσσερις αυτές χώρες. Βλέπουμε ότι η δυσπιστία αυτή υποχωρεί. Έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών του Μαλή, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την Αλγερία και θέλει να δημιουργήσει κάποιες συνθήκες εμπιστοσύνης με τη χώρα αυτή. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες πολύ θετικέ ε, εξελίξεις. Προσπαθήσαμε επίσης να δημιουργήσουμε το ΣΕΜΟΠ, ένα γενικό επιτελείου στρατού, προκειμένου να υπάρχουν κάποιες κοινέ στρατιωτικές επιχειρήσεις και το ΕΦΕΛ, το οποίο αποτελεί ε, μια κοινή προσπάθεια συλλογής πληροφοριών για την περιοχή του Σαχέλ. Το θέμα τώρα είναι να δούμε αν οι πρωτοβουλίες αυτές θα λειτουργήσουν επί τόπου. Θεωρητικά έχουν τεθεί όλες οι βάσεις. Στο Ταμαρασέτ έχει αποφασιστεί να δημιουργηθεί αυτό το γενικό επιτελείο, αλλά δεν έχουμε ακόμα κάποιες συγκεκριμένε στρατικές επιχειρήσεις επιτόπου. Η Μαυριτανοί ήταν αυτή η οποία ήταν έτοιμη να κινητοποιήσει στρατιωτικέ δυνάμει σε συνεργασία με το Μαλί, αλλά δεν έχει ακόμα συντονιστεί από το Ταμαρασέτ. Στόχο μα, στόχο Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζουμε ότι το ζήτημα αυτό θα συζητηθεί σε 15 μέρε όταν οι τέσσερι Υπουργοί Εξωτερικών των ε, κρατών μελών του ΣΟΛΤ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες, παρουσία της κυρίας Άστον και ελπίζουμε ότι τότε θα δοθεί και μια μεγαλύτερη δυνατότητα να εξηγήσουν και τη στρατηγική τους και ελπίζω ότι θα έρθουν και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το πράξουν αυτό. Ελπίζω λοιπόν να τους πείσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει το ΣΕΜΟΠ μέσω του κοινού αυτού Γενικού Επιτελείου Στρατού ότι θα μπορέσει δηλαδή το επιτελείο αυτό όντως να είναι αποτελεσματικό στην πράξη. Οι τέσσερις αυτές λοιπόν χώρες, αντιμετωπίζοντας την αυξανόμενη αυτή απειλή, αποφάσισαν να αυξήσουν τη συνεργασία τους στο Τσάτ, στο Μπουρκίνα Φασό, στη Σενεγάλη και στην Ιγυρία. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό και σε λίγο θα σας αναπτύξω και τη δικιά μου επίσκεψη στην Ιγυρία. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να επεκταθεί η συνεργασία αυτή πέρα από τις τέσσερις αυτές χώρες. Επίσης, στην Αλγερία στις 16 και 17 Νοεμβρίου έλαβε χώρα μία συνάντηση του Παγκόσμιου Φόρουμ κατά της τρομοκρατίας που ουσιαστικά κινητοποίησε το φόρουμ αυτό η κυρία Κλίντον και ήταν παρούσα και η κυρία Άστον. Πρόκειται για ένα φόρουμ το οποίο επικεντρώνεται στο ζήτημα της τρομοκρατίας, αναφέρεται στη στρατηγική του Σαχέλ και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον όμως γιατί απαρτίζεται από 29 κράτη σύν την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχουν πολλά κράτη τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν τρομοκρατία, πολλά μουσουλμανικά κράτη. Πρόκειται δηλαδή για ένα φόρουμ το οποίο ξεκίνησε από το G8 και το οποίο έγινε στη συνέχεια, διευρύνθηκε, όπως ακριβώς και το G8 έγινε G20. Το σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι όλοι οι παράγοντες του Σαχέλ συμμετέχουν. Η Εφρακανική Ένωση, η ΣΕΝΤΕΟ, η μεταβατική κυβέρνηση της Σομαλίας ε, συμμετέχει το Μαρόκο, το Μαλί και πολλές άλλες χώρες της περιοχής του Σαχέλ. Πρόκειται λοιπόν για μια σημαντική πρωτοβουλία, για ένα φόρουμ το οποίο πρόκειται να επεκταθεί ακόμα περισσότερο και να οδηγήσει σε συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένες επιτρόπου δράσης. Επίσης, μια άλλη πρωτοβουλία, για την οποία δεν υπάρχει ακόμα απόλυτη συνένεση από όλους, θέλουμε να καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε την συνεργασία μας για ζητήματα άμυνας, προκειμένου να καταφέρουμε να υποστηρίξουμε περισσότερο τη στρατηγική που έχουμε για το Σαχέλ. Πρόκειται μια πρωτοβουλία που ακόμα εξετάζεται, δεν έχουμε ακόμα την έγκριση της ύπατη εκπροσώπου. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο θα εξεταστεί ακόμα περισσότερο από τα 27 κράτη της ε, Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Θέλουμε να καταφέρουμε να έχουμε μια ελαφριά συνεργασία, μη στρατιωτική, ενδεχομένως στο Βόρειο Νίγηρα καταρχάς, είναι πάντως μια πρωτοβουλία την οποία ακόμα εξετάζουμε. Και τρίτη και τελευταία εξέλιξη όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ιγυρία αυτή τη φορά. Ήμουν εκεί την προηγούμενη εβδομάδα με τον συντονιστή του Σαχέλ και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε καλύτερα πώς εξελίσσεται η πολιτική κατάσταση στη χώρα και ποια είναι η πολιτική τη Νιγηρίας. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να πω ότι έχω μια απόλυτα ξεκάθαρη κατάσταση όσον αφορά τις ε, τρομοκρατικές ομάδες που αναπτύσσονται στην χώρα αυτή. Δεν ξέρουμε αν πρόκειται για ομάδες που έχουν μια τοπική ατζέντα και που σιγά σιγά θα γίνουν παρακλάδι της Αλκάιντα ή αν πρόκειται για ένα συνονθήλευμα εγκληματικών κινημάτων με κάποια πολιτική διάσταση. Τα πράγματα παραμένουν ακόμα αρκετά σαφή. Πρόκειται πάντως για ένα κίνημα το οποίο είναι περιορισμένο ακόμα, δεν έχει πολλά μέλη, αλλά μπορεί ενδεχομένως να διευρυνθεί, να απτυχθεί ακόμα περισσότερο. Ακριβώς επειδή οι δυνατότητες στρατολόγησης είναι πάρα πολύ σημαντικές στο βόρειο Νίγηρα. Υπάρχουν πολλοί νέοι, νέα παιδιά ουσιαστικά, τα οποία εγκαταλείπουν τις οικογένειές τους ουσιαστικά στρατολογούνται από τις ομάδες αυτές, από την ομάδα Boko Haram. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό έχει πολλές αρνητικές συνέπειες. Η συνεργασία των υπηρεσιών του στρατού, των υπηρεσιών πληροφοριών, των αστυνομικών υπηρεσιών θα πρέπει να ενταθούν προκειμένου να ανταποκριθούμε στην απειλή αυτή της τρομοκρατίας. Οι ε, αρμόδιες αρχές ε, της χώρας με τους οποίους ε, συναντηθήκαμε θέλουν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ανάπτυξη και την ασφάλεια. Στα πλαίσια της αναπτυξιακής μας πολιτικής για την Νιγηρία, μέχρι στιγμής είχαμε επικεντρωθεί στις αποσχιστικές αυτές δυνάμεις που είχαμε δει και που συνδέονται με την εκμετάλλευση του πετρελαίου και βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα κάποια προβλήματα πειρατείας. Αυτά ήταν τα ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο χριστιανικό νότο της χώρας. Βλέπουμε όμως τώρα ότι η χώρα απαιτεί μια κάποια υποστήριξη προκειμένου να απτυχθεί και το βόρειο τμήμα της και θα πρέπει βέβαια να υπάρχει σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΥΠΑ της εκπροσώπου και θα πρέπει να εξορροπήσουμε τη συνεργασία που έχουμε με την Ιγυρία προκειμένου να καταφέρουμε να βοηθήσουμε όχι μόνο τον Νότο αλλά και το Βορρά της χώρας για την ανάπτυξη και την ασφάλεια. Η στρατηγική λοιπόν του Σαχέλ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Θα πρέπει να διαμορφωθεί, να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες. Οφείλουμε να είμαστε παρόντες στο Σαχέλ θα πρέπει να προλάβουμε την ε, ανάπτυξη της τρομοκρατικής αυτής απειλής στο Σαχέλ, προτού αυτή αναπτυχθεί εντελώς. Αυτά είχα να σας πω εν είδη Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση, όπως πάντα πολύ σαφής, ε, όχι κατά ανάγκη καθησυχαστική φυσικά. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πάντα δύσκολο να ακολουθήσεις τον Ζιλντοκιακόφ, γιατί καλύπτει ε, υπέροχα όλες τις πτυχές. Θα ήθελα να προσθέσω κάποια σημεία κι εγώ με τη σειρά μου. Πρώτα απ' όλα δεν πιστεύω ότι είναι αναγκαίο εδώ να επενθυμίσουμε τους τέσσερις άξονες της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασφάλειας και Ανάπτυξης στο Σαχέλ. Ε, πρώτα απ' όλα γιατί έχουν ήδη αναφερθεί από τον προλαλήσαντα και ε, νομίζω είχατε ήδη μια συζήτηση μόλις προηγουμένως. Θα ήθελα να φυσίσω την προσοχή σε ένα σημείο που δεν αναφέρθηκε όμως, το θέμα της πρόληψης της ε, βίαιης ριζαστικοποίησης, που είναι μία από τις συνιστώσεις της στρατηγικής και που είναι ένα σημαντικό μέρος, διότι υπάρχουν φαινόμενα προσιλητισμού ε, που σχετίζονται με θέματα είτε ε, προηγουμένων ε, ανταρτικών ομάδων ή σε σχέση με συζητήσεις που αφορούν το Ισλάμ, άρα είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από διευθετήσεις που θα πρέπει να προσδιοριστούν και να μελετηθούν μέσα από μη κρατικούς ε, παίκτες, να δούμε πώς μπορούμε να ε, αντιταχθούμε σε αυτό το, τη ριζοστικοποίηση. Είναι αλφές ότι ε, από τότε που ξεκίνησε η στρατηγική σταθερότητα και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε θετικές επιπτώσεις αφενός ε, στην τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον στην παγκόσμια αρένα ε, στο θέμα των προκλήσεων του Σαχέλ. Η προσέγγιση μας αναγνωρίζεται από τις χώρες εταίρους της περιφέρειας αλλά και από άλλες ε, ε, χώρες παγκοσμίω, ως μια στρατηγική που είναι επαρκώς ανοιχτή στα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν και που έχει ε, δυνατά σημεία σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την ανάπτυξη, αλλά και σε άλλους τομείς. Από τη μια πλευρά, λοιπόν, έχουμε τοποθετηθεί σωστά στο πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις απειλές. Από την άλλη πλευρά, ε, μια καλύτερη δυναμική ε, σε ό,τι αφορά τις χώρες που αντιμετωπίζουν τις απειλές ε, και την συνεργασία τους. Αυτό το έχουμε ήδη ακούσει για την διάσκεψη στο Αλγέρι, το νέο πλαίσιο του Παγκοσμίου Φόρουμ. Όλα αυτά είναι εξελίξεις πολύ ενθαρρυντικές κατά την άποψή μου. Αυτό που ίσως θα έπρεπε να ξαναδούμε είναι ότι παραμένουν κάποιες δυσκολίες στο διάλογο και τη συνεργασία ανάμεσα στις ε, άμεσα εμπλεκόμενες χώρες. Η κριτική που ακούγεται πολύ συχνά είναι ε, απέναντι στο Μαλί ε, σε ό,τι αφορά την αντίδραση που απαιτείται από κάποια χώρα στην επικράτεια της οποίας βλέπουμε να αναπτύσσονται τρομοκρατικές ομάδες όπως αυτές της ΑΚΜΗ αλλά έχουμε την κριτική απέναντι στο Μαλί και στο Νίγηρα, απέναντι στην Αλγερία, διότι η Αλγερία ε, κρατάει κάπως τον ηγετικό ρόλο στην περιοχή και δεν βλέπουμε την συνεργασία ανάμεσα στις χώρες αυτές. Ε, θα μπορούσα να σας ε, αναφερθώ και στην επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα μαζί με τον Επίτροπο Πίμπαλς. Ε, βλέπουμε μια πολιτική βουλσιαρχία και στρατιωτική από πλευράς κάποιων χωρών που είναι αξιοσημείωτη. Άρα έχουμε ακόμη να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα της διαφορετικής εκτίμησης των δεσμεύσεων. Έχω γνωρίζουμε και ε, τα παράπονα του Πρόεδρου Αζής της Μαυριτανία που πιστεύει ότι η χώρα του καταβάλει πολλές προσπάθειες αλλά οι προσπάθειες αυτές δεν αναγνωρίζονται πάντα. Πιστεύω ότι έχουμε θετικές εξελίξεις, έχουμε ακόμη προκλήσεις ό,τι αφορά την περιφερειακή συνεργασία Ίσως ε, να υπάρχει μια άλλη διάσταση, αποσύνδεση ανάμεσα στο πολιτικό και το τεχνικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο, ένα παράδειγμα, είναι οι τέσσερις Υπουργοί Εξωτερικών που προσέρχονται στην Βρυξέλλες, που ήταν στην Ουάσιγκτον και που επιδεικνύουν την πολιτική βούληση των τεσσάρων χωρών εμπλεκομένων χωρών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ασφάλειας και ανάπτυξης ε, στο Σαχέλ και επίσης η μετάφρασή τους στη συνεργασία επιτόπου ε, σε ό,τι αφορά το ε, κέντρο των Γενικών Επιτελείων ΣΑΤΟΥ. Βέβαια, εκεί Μέχρι στιγμής δεν είδαμε συγκεκριμένη συντονισμένη δράση επιτόπου. Οι ομάδες έχουν περιορισμούς όπως γλωσσικούς ε, περιορισμούς. Έχουμε τους αραβόφωνες και τους γαλλόφωνους. Ε, όταν πρόκειται για συντονισμό δράσεων, αντιμετώπισαν αυτό το φραγμό, το γλωσσικό φραγμό, στον οποίο δεν έχουν ακόμη βρεθεί όλες οι λύσεις. Άρα, υπάρχει μια αποσύνδεση ανάμεσα στην πολιτική βούληση και την βούληση πραγματικής συνεργασίας επιτόπου. Βέβαια, ε, θα μπορούσαμε εμείς να συνεισφέρουμε, ίσως με την προώθηση του ε, κολεγίου ε, συνεργασίας στο ΣΑΧΕΛ, θα μπορούσε να, ε, να συνεργαστεί με τα γενικά επιτελεία ή να κάνουμε μία ειδική αποστολή στήριξης του συντονισμού αυτών των γενικών επιτελείων. Ε, νομίζω βλέπουμε και μία διεύρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες. Ο Ζιλ το έχει αναφέρει. Ε, σε επίπεδο σε ΜΟΚ οι, χώρες παραμένουν το, Αλγέρι, το Μάλι, η Μαυριτανία και ο Νίγηρας. Υπάρχει συνεργασία. Έχουν ήδη κληθεί να έχουν προσκαλέσει άλλες χώρες όπως το Μπουρκίνα, Φασό, το Τσάντ, την Ιγυρία και μια άλλη χώρα χώρα που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή ίσως στη Σενεγάλη. Έχουν καλέσει αυτές τις χώρες να συμμετέχουν και βλέπουμε μια διεύρυνση της συνεργασίας και αυτό είναι θετικό, ένα θετικό βήμα διότι ε, υπάρχουν δεσμοί που αρχίζουν να δημιουργούνται και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στο επίπεδο Τη υλοποίηση της στρατηγική στο Σαχέλ. Πιστεύω ότι θα μπορούμε να είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι με το τι ξεκίνησε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στην ε, ανάπτυξη, όπως αναφέρθηκε ήδη. Έχουμε πρόσθετους σπόρους που δόθηκαν στο Μαλί και στο Νίγηρα που έχουν υπογραφεί στο Μπαμακό, στην Παμακό και στην ΙΑΜΕΙ από τον Επίτροπο Πίπαλς. Είναι κονδύλια τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα σε ορισμένες δράσεις δέσμευσης στον τομέα της δικαιοσύνης ή το τομέα της ε, ανάπτυξης ε, δυνάμεων ασφάλειας, κρατικής ασφάλειας στο Μάλι. Ε, ήδη είμαστε στην επιχειρησιακή φάση για κάποιες συνιστώσεις αυτών των επιπροσθέτων κονδυλίων. Αυτά τα επιπρόσθετα κονδύλια ε, δόθηκαν επίσημα στις χώρες αυτές και θα χρηματοδοτήσουν δράσεις ε, για τον απεγκλωβισμό ε, ζωνών που είναι ιδιαίτερα μη προσπελάσιμες στο Βόρειο Νίγηρα ή στο Βόρειο Μαλί και στήριξη στον τομέα της δικαιοσύνης, στον τομέα της ασφάλειας, πολιτικής ασφάλειας και σε δράσεις και διαδράσεις με την κοινωνία των πολιτών, είτε για την προώθηση ε, δραστηριοτήτων που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, είτε στο τομέα της ε, μάχης κατά της ρίζοσπαστικοποίησης. Εάν η υλοποίηση ε, μέσα από τα κονδύλια του ε, Ταμείου και μέσα από αυτά που ανέφερε ο Ζιλ, αν αυτά δείχνουν μια σωστή αντίδραση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως ε, να μένει ακόμη δουλειά να γίνει σε ό,τι αφορά τα ε, μέτρα ε, στήριξης στον τομέα της ασφάλειας. Ξεκινούν οι συζητήσεις για μια αποστολή στον Νίγηρα βέβαια εάν τα κράτη-μέλη θα συμφωνήσουν για αυτή την αποστολή που θα συζητηθεί ε, λίαν συντόμως. Ε, Θα έλεγα επίσης ότι ο Πίτροπος Πίμπαλ όπως γνωρίζετε πολύ καλά, χειρίζεται τα ταμεία ανάπτυξης και ε, επιθυμεί πάρα πολύ όπως αυτά τα κονδύλια να μην χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Σε πάση περιπτώσει παρατήρησε στην ε, επίσκεψή του αυτή την καθυστέρηση ε, στον τομέα της ασφάλειας και τον ενδιαφέρε να δει εάν μέσα από το African Peace Facility που είναι ένα από τα ταμεία που συν, τη συνδιαχείρισης θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε το Μάλι και τον Νίγηρα. Ίσως να πω κάτι για τους κινδύνους διασύνδεσης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ο Γιώργος Κέρκοφ αναφέρθηκε στους πιθανούς κινδύνους ανάμεσα στα μονάδες ΑΚΜΗ και ΜΠΟΑΚΜΑ. Ε, μια χώρα όπως ο Νίγηρας αντιμετωπίζει και γεωγραφικά αυτό το πρόβλημα, διότι έχουν την ακμή στο βορρά και τους κινδύνους από την Μποκοχαράμα στον νότο και ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες ασφάλειας αυτών των χωρών είναι πεπισμένες ότι έχουν ε, αποδείξεις ότι υπάρχουν επιχειρησιακοί δεσμοί ανάμεσα στις οργανώσεις αυτής. Ε, πρέπει βέβαια να ληφθούν όλες οι, όλα τα μέτρα προστασίας. Βέβαια υπάρχουν αυτές οι διασυνδέσεις και μπορεί να αναπτυχθούν και είναι σημαντικό πως η στατική του Σαχέλ και των χωρών που εμπλέκονται να παρακολουθούν την κατάσταση στο Βόρειο ε, Νίγηρα ε, σε συνεργασία με την Νιγηρία, που είναι πολύ σημαντική. Να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόγραμμα συνεργασίας με την Νιγηρία δεν είναι τόσο στοχευμένο ε, στο νότο ως ως όσο στο βορρά. Ε, υπάρχουν, ε, υπάρχει υποστήριξη στα, στα κράτη του βορρά που έχουν αποτελέσματα στο τομέα της εξυγίανσης, αλλά σε ό,τι φορά την στήριξη, πρόληψη συγκρούσεων και εντάσεων, αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή στον Ήγηρα και θα πρέπει να ενισχυθεί και στο Βορρά όπου υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και προκλήσεις ε, ανέχειας ε, και εντάσεων ε, εθνικών, θρησκευτικών και με παρακλάδια τρομοκρατικά αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Κάτι άλλο το οποίο δεν είναι διασύνδεση ανάμεσα σε οργανισμούς, αλλά είναι ένα άλλο πρόβλημα, το πρόβλημα της μη ασφάλειας και ε, λόγω της παράνομης διακίνησης ε, στο ΣΑΚΕΛ και της παράνομης διακίνησης και ε, ένα ξεκίνημα πειρατείας στον κόλπο της Γουινέας. Χώρες όπως η Νιγηρία αντιμετωπίζουν και τα δύο φαινόμενα και είναι σημαντικό στην στο όραμά μας για να αντιμετωπίσουμε και τα δύο προβλήματα, να έχουμε αυτό κατά νου για να προσαρμόσουμε τη στρατηγική μας και τους διάφορους τρόπους παρέμβασης. Και είναι σημαντικό το επίπεδο επέμβαση των περιφερειακών οργανώσεων. Ο Επίτροπος Λαμάμρα ήταν εδώ πριν από λίγο. Για την ώρα η εμπλοκή της, Ευρω... Αφρικανικής Ένωσης, της ECOWAS, στα προβλήματα του Σαχέλ είναι ε, πενιχρή. Ε, χρειάζεται να διπλασιάσουμε τις προσπάθειες αυτών, έτσι ώστε αυτές οι οργανώσεις να συνεισφέρουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ε, ασφάλεια στον κόλπο της ε, Γουινέας, ε, βλέπουμε την οργάνωση της Κεντρικής Αφρικής της ΕΜΑΚ που έχουν υλοποιήσει δράση συντονισμού περιπολιών της ακτοφυλακής εδώ λοιπόν πρέπει να συνεισφέρει ακόμη περισσότερο αυτή η οργάνωση. Ε, κάτι άλλο σχετικά με την επίσκεψη των τεσσάρων υπουργών της Αλγερίας, του Νίγηρα και της Μαυριτανίας. Προβλέπεται να γίνει στι 8 Δεκεμβρίου. Εάν το Κοινοβούλιο ε, ε, θα θέλαμε να ακούσουμε και από το Κοινοβούλιο γιατί 8 ή 9 Δεκεμβρίου θα πρέπει να προτείνουμε κάτι αλλιώς θα υπάρχει μια άλλη ευκαιρία. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο στις 8 και 9, 8 του μηνό είναι πέμπτη. Μου φαίνεται λίγο πολύπλοκο πάντως. Ε, σας ευχαριστώ πολύ πάντως που μας το λέτε, γιατί θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε και εμείς τους τέσσερις υπουργούς σε σχέση με τα όσα είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί ε, μας είπατε ότι επιταχύνεται η στρατηγική του Σαχέλ και ότι είναι ικανοποιητική όσον αφορά την πτυχή της στην αναπτυξιακή. Σας υπενθυμίσω και το πάλωστε και ο κύριος Ντεκέρκοφ ότι ε, υπάρχει μία δυσκολία όσον αφορά την πτυχή ασφάλειας. Το ζήτημα είναι σαφώς πιο ευαίσθητο, πιο λεπτό Πρέπει προφανώς να γίνει μια διαπραγμάτευση με τις εμπλεκόμενες χώρες, αλλά γιατί υπάρχουν και δομές της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν βοηθούν πάρα πολύ την ε, σφαιρική αυτή προσέγγιση. Πολλές φορές ε, στα πλαίσια μιας σφαιρικής προσέγγισης αποδυναμώνεται περισσότερο η πτυχή της ασφάλειας, ιδίως όταν θέλουμε να έχουμε μια κρατεά ασφάλεια, hard security. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια της στρατηγικής του Σαχέλ να έχουμε και τις δύο πτυχές, και την πτυχή της ανάπτυξης και την πτυχή της ασφάλειας. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εντάξουμε και την κοινή εξωτερική πολιτική ασφάλειας και άμυνας στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε τα μέσα τα οποία προβλέπονται στα πλαίσια της στρατηγικής του Σαχέλ και ενδεχομένως και κάπως ηρωνικά θα μπορούσε να πω και το ακόλουθο. Το είδαμε και στη Λιβύη. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει όλες ε, οι δομές του ΕΚΟΑΣ να αναλάβουν τις ευθύνες τους μέχρι το πιο υψηλό επίπεδο, γιατί πολύ συχνά βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι δισταγμοί απέναντι στην κοινή εξωτερική πολιτική ασφάλειας και άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι προέρχονται από τις ίδιες τις ε, χώρες ε, ΕΚΟΑΣ. Πολλούς δισταγμούς επίσης έχουμε και από τα κράτη-μέλη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής να κινητοποιηθούν όλες οι δομές και να έχουμε και τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και γενικότερα τη συνεργασία των δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνω λοιπόν την έκκληση αυτή γιατί δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί μια κατάσταση σε αυτή της Λιβύης όπου πολλές φορές ήμασταν κάπως εξωτερικοί παρατηρητές στην όλη υπόθεση. Η κυρία Γκόμες θέλει το λόγο πρώτα. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπατε κύριε Πρόεδρε. Και εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και συγκεκριμένα η κυρία Άστον θα πρέπει να εντατικοποιήσει την διαδικασία αυτή και να καλέσει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Μιλάμε ουσιαστικά για την πίσω αυλή μας εδώ, για την άμεση γειτονιά μας. Ουσιαστικά τίθεται να αφιβόλω η ίδια η δική μας η ασφάλεια και βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες ε, πιέσεις όσον αφορά τους ε, αμυντικούς προπολογισμού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή επιμέρους τα κράτη-μέλη πιέζονται δημοσιονομικά, είναι πολύ σημαντικό να συστρατεύσουμε τις δυνάμεις μας, από κοινού να κινηθούμε. Και ιδίω όσον αφορά για μια αποστολή της ΚΕΠΑ, είτε πρόκειται για τη Λιβύη, είτε πρόκειται για την εφαρμογή της στρατηγικής του Σαχέλ. Πέραν των όσων θα κάνουμε στη Λιβύη δηλαδή, όσον αφορά το ζήτημα αυτό, ενδεχομένως η σκληρή αυτή ασφάλεια να είναι απαραίτητη, όπως είπατε, αλλά ενδεχομένως η σκληρή αυτή διάσταση, η διάσταση hard στην οποία αναφερθήκατε, να έρθει τελικά από του ίδιου ανθρώπινου πόρου, από την ίδια την ανθρώπινη πυρογνωμοσύνη, από τις πληροφορίε που θα έχουμε. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση πάντως να δραστηριοποιηθούμε το συντομότερο δυνατό. Και έχω και ένα ερώτημα. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε μία αποστολή ΚΕΠΑ Σαχέλ η οποία να εμπεριέχει τις αρμοδιότητες που θα έχουμε και στην ε, Λιβύη ε, σε συνεργασία πάντα με, τις, με τα Ηνωμένα Έθνη και με τον καταμερισμό των ε, αρμοδιοτήτων και σε συνεργασία βέβαια με τις αρχές της Λιβύης ή θα έχουμε μία αποστολή ΚΕΠΑ Λιβύη ξεχωριστή από τη στρατηγική που θα έχουμε στο Σαχέλ, από την αποστολή που θα έχουμε στο Σαχέλ. Και η αποστολή στη Λιβύη στην περίπτωση αυτή θα υποστηρίζει κυρίως ε, την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων και θα ασχοληθεί επίσης και με το ζήτημα του αφοπλισμού και με την ε, μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας. Και ένα ερώτημα ακόμα. Από όσο κατάλαβα, πριν από έναν ή δύο μήνες, γύρω στο Σεπτέμβριο, τα όσα συμφωνήσαμε στη διάσκεψη των Παρισίων ήταν τελικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθούσε να ταυτοποιήσει να εντοπίσει τις ανάγκες στο ζήτημα αυτό της ασφάλειας των συνόρων κτλ. Αλλά δεν είχε αποφασιστεί ακόμα τότε ποιος θα αναλάμβανε το ρόλο αυτό της υποστήριξης των λιβικών δυνάμεων. Καταφέραμε να ξεπεράσουμε το ζήτημα αυτό, βρισκόμαστε πλέον σε μια νέα φάση όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Και κάτι ακόμα το οποίο θέλω να σας ρωτήσω. Όσον αφορά την Αλγερία. Κοιτάξτε, εγώ ανησυχώ ιδιαίτερα. Αναφερθήκατε εσείς σε κάποιες θετικές εξελίξεις στη χώρα αυτή. Είπατε ότι η Αλγερία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για μια περαιτέρω συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συντονισμό με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Ωστόσο, έχω το ακόλουθο ερώτημα. Είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Ποια είναι η δική σας αξιολόγηση όσον αφορά την κατάσταση της Αλγερίας, γιατί δεν ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμη στο παρελθόν, ιδίως κατά τη διάρκεια της κρίσης στη Λιβύη. Το αντίθετο μάλιστα. Όντας στη Λιβύη, άκουσα πολλούς πολίτες οι οποίοι θεωρούσαν ότι η Αλγερία συνεργαζόταν με το αντίπαλο στρατόπεδο ουσιαστικά. Υποστήριζε ότι είχε απομείνει από το καθεστώς Καντάφη όσο βρισκόταν εκεί. Και στο Σαχέλ έχουμε και πάλι εκεί ένα συγκεκριμένο ρόλο της Αλγερίας και συγκεκριμένες πιέσεις που είχε ασκήσει το καθεστώς της Αλγερίας. Ποια είναι λοιπόν η δική σας άποψη σε σχέση με όλα αυτά. Ποια θα είναι η θέση της Αλγερίας και η στάση της σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Και κάτι ακόμα. Γνωρίζουμε ότι στη Λιβύη προφανώς κυκλοφορούσαν ε, παντός ειδός ε, όπλα. Κατά τη διάρκεια όμως της ε, καταπολέμησης του καθεστώτος ε, του Καντάφη προστέθηκαν ακόμα περισσότερα όπλα τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί και από το Κατάρ. Όχι επίσημα ενδεχομένω από το κράτος του Κατάρ, αλλά από κάποιες αρχές σημαντικές μπορούμε να πούμε της χώρα αυτής. Και προφανώς τα όπλα αυτά είναι αυτά τα οποία τελικά κατέληξαν στα χέρια των συντηρητικών Ισλαμικών ε, Λιβικών δυνάμεων που δεν συνδέονται απαραίτητα με την Αλκάιντα, αλλά έχουν κάποιες φονταμεταλιστικές θρησκευτικέ προτερότητες, μια φονταμελιστική ατζέντα. Διερωτώ με λοιπόν, η ενίσχυση αυτή όλων αυτών των φονταμεταλιστικών κινημάτων που μπορεί να έχουν σχέσεις με την Αλκάιντα ή που συνδέονται με τον Μποκοχαράμ στην Βόρεια Νιγηρία, από πού προέρχεται η χρηματοδότησή τους. Γιατί πέρα από τους κινητήρους βασικούς λόγους, πέρα από, τις, από τη στρατολόγηση αυτή, πρέπει κανείς να έχει και χρήματα προκειμένου να διεξάγει αυτές τις δραστηριότητες. Σας ευχαριστούμε κυρία Νικολάη. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, αλλά θεωρώ αυτό το θέμα μία από ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για το ζήτημα της ασφάλειας. Το 2010 από τη στρατηγική ασφάλειας είχαμε τις μεγάλες αλλαγές ε, του τοπίου στη Βόρεια Αφρική. Και Γι' αυτό χρειαζόμαστε πιο ισχυρές ε, λύσεις για την περιοχή αυτή. Αν συγκρίνεται με την κατάσταση στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν, δεν έχει αλλάξει τίποτα στον αφορά την Αλκαΐντα ε, σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Είναι μια πάρα πολύ γόνιμη περιοχή για τομοκρατικές ενέργειες και οργανώσεις διότι υπάρχει ψηλό επίπεδο φτώχειας και ανασφάλειας και επίσης ε, πάρα πολύ μεγάλη διαφθορά. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν τη γνώμη σας ε, σε σχέση με τη διαφθορά σε κρατικό επίπεδο. Ε, αυτό που μας καίει ιδιαίτερα είναι η τρέχουσα κατάσταση στη Λιβύη. Δυστυχώς ο Καντάφη είχε προσλάβει μισθοφόρους κυρίως από το Τσάντ. Ε, θυμόσαστε τι είχε συμβεί το, στο Ιράκ με τον Σαντάμ Χουσέιν πολλοί ε, πρώην ε, στρατιώτες της άναπλες δυνάμεις του Ιράκ έχουν μετακινηθεί προς τα εκεί. Πιστεύετε ότι αυτές οι στρατιωτικές δυνάμεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα τέτοιο είδους οργάνωση, διότι μπορεί ενδεχομένως όλοι αυτοί οι μισθοφόροι, οι πρώην στρατιώτες κλπ. να οδηγήσουν στην επιδείνωση της κατάστασης ε, ασφάλειας, διότι είναι πολύ δύσκολο δύσκολο να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στη Βόρειο Αφρική ε, γενικά για όλη την περιφέρεια από πόψεως ασφάλειας, διότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το πολιτικό μέλλον η Λιβύη μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στις όμορες χώρες. Οι ορισμένοι στη Λιβύη ζητάνε την επιβολή του Ισλαμικού νόμου, Σαρία. Υπάρχουν παρόμοια αιτήματα και κινήματα που ακούγονται στην Αίγυπτο. Λοιπόν, ε, είναι πολύ σοβαρό το θέμα διότι θα έχει επιπτώσεις. Και η τελευταία ερώτηση. Πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική που είναι γενικής φύσεως πρέπει να εκπροσωπεί την ε, γενική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καιρούς ειρήνης. Όμως τώρα δεν είμαστε σε καιρούς ειρήνης και αυτή η πολιτική ευρωπαϊκή θα πρέπει να αναβασμιστεί με συγκεκριμένα μέτρα ε, σήμερα και με συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση διότι πιστεύω ότι τα μέτρα τα οικονομικά τα οποία προβλέπονται σήμερα δεν είναι αρκετά με τα νέα δεδομένα. Ευχαριστούμε καταρχάς ο κύριος Δεκέρκοφ. Όσον αφορά την ερώτηση της κυρίας Γκομές, ξεχωριστή ή κοινή αποστολή. Εγώ θα έλεγα ξεχωριστή, γιατί διαφορετικά είναι τα προβλήματα της Λιβύης άλλη στάση στο Σαχέλ. Εγώ πάντα έλεγα ότι θα έπρεπε να είχαμε μια αποστολή ΚΕΠΑ στο Σαχέλ, προκειμένου να καταφέρουμε να αποκρισταλώσουμε την πολιτική βούλησή μας. Με δύο τρόπους θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ορισμένοι θεωρούν ότι επειδή έχει διαφορετική στάση το Μαλή θα πρέπει να καταφέρουμε να ενισχύσουμε την Ιγυρία και το... τη Μαυριτανία. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη παρουσία οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονε και κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε περισσότερου πόρου και να έχουμε και διμερεί ε, συνεργασίε. Ισπανία, Γαλλία και άλλε χώρε ε, είναι παρούσες ε, όσον αφορά τις υποδομές, όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα. Η μεγαλύτερη λοιπόν πρόκληση είναι η πολιτική βούληση και ο συντονισμός λοιπόν. Θα επιθυμούσα να καταφέρουμε και στα κράτη-μέλη και στην ΕΚΟΑΣ να υπάρχει απαραίτητη συνένεση. Συμφωνώ πάντως μαζί σας. Όντως, ε, ο χαρακτήρας είναι κατεπήγον και πρέπει να κινητοποιηθούν επιγόντως ε, τα μέσα. Δεν παρακολουθώ εκ του σύνεγγυ το ζήτημα της Λιβύης, επομένως θα ήμουν αρκετά προσεκτικό στα σχόλια τα οποία θα κάνω. Πάντως, ε, ακόμα βρισκόμαστε στη φάση του εντοπισμού των αγκών στα πλαίσια της απόφασης επιμερισμού που ελήφθη στο Παρίσι, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε την, τον εντοπισμό των αγκών όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων, όσον αφορά την κοινωνία των πολιτών και όσον αφορά την, ε, τη δημόσια επικοινωνία. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρηγορότερα. Μία δυσκολία που αντιμετωπίζουμε είναι ότι δεν έχουμε ακόμα τις ε, αντίστοιχες ε, δυνάμεις, τις αντίστοιχες αρχές από πλευράς Λιβύης. Αυτή τη στιγμή διοργανώνεται το Λιβικό κράτος Πάντως ε, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι μας δόθηκε ως αρμοδιότητα η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Έχουμε πυρογνωμοσύνη στο ζήτημα αυτό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα, ιδίως όσον αφορά τη δραστηριότητα του αφοπλισμού και θα πρέπει να είμαστε κάπως προδραστικοί, προορατικοί ως προς αυτό. Όσον αφορά τώρα την Αλγερία, είναι σαφές ότι έχει αλλάξει η στάση πλέον της χώρας αυτής. Δεν είναι μυστικό αυτό. Και αυτό προφανώς οφείλεται στο ότι από τη μια έχουμε την Αραβική Άνοιξη που αλλάζει πλέον τα δεδομένα για το σύνολο της όχθης αυτής της Μεσογείου και από την άλλη έχουμε και μια πιο προσεκτική στάση από πλευρά Αλγερινών αρχών όσον αφορά τη λιβική κρίση. Θεωρεί λοιπόν η Αλγερία ότι έχει έρθει κατάλληλη στιγμή να βγει από τον αποκλεισμό της και να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα. Πάντως δεν έχω λόγο να θέτω να αμφιβόλω την ειλικρίνεια των προθέσεων αυτών, πάντως θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί η πρόοδος, προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα πραγματικό πολυμερικό χαρακτήρα των, της συνεργασίας της χώρας αυτής με τα κράτη του Σαχέλ. Θα πρέπει η χώρα να συνεχίσει να κινείται στην οδό αυτή και αυτό αποτελεί πρόκληση βέβαια και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα πρέπει να δημιουργήσει μια ε, απτή συνεργασία με την Αλγερία. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή, αλλά θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε ανώτατο επίπεδο. Η συνεργασία μεταξύ Γαλλία και Αλγερία, για παράδειγμα. Πήγα στην Αλγερία πρόσφατα, το, το Σεπτέμβριο και τον Ιούνιο, και βλέπω ότι η κατάσταση έχει πλέον βελτιωθεί. Ο Υπουργό Εξωτερικών τη Γαλλία, κ. Ζουπέ, πήγε στην Αλγερία και υπάρχει πλέον ένα πολύ πιο θετικό και φιλικό κλίμα. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνει η κατάσταση αυτή ακόμα πιο απτή, ακόμα πιο ρεαλιστική και το ΣΕΜΟΚ θα πρέπει να γίνει κάτι το πολύ πιο απτό και συγκεκριμένο. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των διαφόρων ομάδων από την Αλκάιντα, συμφωνώ ότι πολύ συχνά μέσω των λίτρων αυτών που ζητούνται από τις απαγωγές ουσιαστικά χρηματοδοτείται η ΑΚΜΗ, η Αλκάιντα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ. Δεν υπάρχει ακόμα μια κοινοτική συνένεση όσον αφορά την δική μας δράση για το ζήτημα αυτό. Όσον αφορά το θέμα της διαφθοράς, Πράγματι, όσον αφορά τη διεθνή κατάταξη διαφάνειας, θα δείτε την άμεση σχέση μεταξύ του προβλήματος ε, και της γεωγραφικής τοποθεσίας αυτών των κρατών. Η διαφθορά είναι ένα σημαντικό συστατικό του όλου προβλήματος. Και για τη Λιβύη και πάλι είμαι επιφυλακτικό όσον αφορά την ε, μετατροπή των μισθοφόρων σε εγκληματίες. Ε, δεχομένως, ε, εντάξει, υπάρχει μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε πρόθεσμα. Σημερίζουμε τις επιφυλάξεις σας. Αυτοί οι άνθρωποι, οι πρώην, μισθοφόροι κλπ. δεν είναι εύκολο να γίνουν ξαφνικά, ας πούμε, κάτι άλλο, επιχειρηματίες, δεν ξέρω εγώ κάτι άλλο. Ελπίζω όμως ε, και δεδομένου ότι συμμερίζουμε την εκτίμησή σας να μπορούν ε, τουλάχιστον όσοι ήταν στις άνοπλες δυνάμεις να παίξουν έναν επικοδομητικό ρόλο στο μέλλον. Για, τις, ε, για το Σαχέλ 400 συν 150 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι αμεληταίο ποσόν. Δεν είναι τόσο πολύ χρηματικό το πρόβλημα, δηλαδή να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και με τους Καναδούς και με τους ε, ε, Αμερικανούς και να συνδυάσουμε τη δεξαμενή οικονομικών πόρων ε, και να ενδεχομένως κινητοποιήσουμε κονδύλια από την Ιαπωνία. Δεν είναι τόσο το θέμα λοιπόν του ποσού, αλλά το πόσο γρήγορα μπορούμε να αντιδράσουμε και πόσο γρήγορα μπορούμε να αναπτύξουμε την πτυχή ασφάλειας της όλης στρατηγικής για την περιοχή. Ευχαριστώ. Στο θέμα του ρόλου ηγεσία τη ΕΔ στο θέμα της ασφάλειας και της ανάπτυξη, νομίζω συμφωνούμε απόλυτα. Στην περίπτωση του Σαχέλ, πιστεύω ότι υπήρξε κάποια καθυστέρηση, που όπως είπε και ο Ζιλ, οφείλεται στην ευαισθησία του θέματος μέρη. Υπάρχουν επιφυλάξεις από τη μια πλευρά να θέσουμε ένστολους εκεί στο Σαχέλ λόγω των επιπτώσεων που μπορεί να έχει, πολιτικών επιπτώσεων και της εικόνας που θα δημιουργηθεί και υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που έχουν και προβλήματα προπολογισμού, όπως γνωρίζετε. Γι' αυτό υπήρξε κάποια καθυστέρηση από πλευρά ΚΕΠΑ στο Σαχέλ αλλά η συζήτηση έχει ξεκινήσει και προχωράει και πιστεύω ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα παίξει τον ρόλο της προωθώντας μία απαραίτητη συνένεση. Συμφωνώ μαζί σας κυρία Γκόμες ότι η, μια αποστολή της ΚΕΠΑ του Σαχέλ ε, θα πρέπει να επικεντρωθεί στα θέματα δυνατοτήτων, ενίσχυσης των ε, ανθρωπίνων πόρων επιτόπου, είτε της αστυνομίας είτε του στρατού και επίσης ε, στο θέμα του εξοπλισμού διότι υστερούν στο θέμα αυτό, ε, εξοπλισμό επικοινωνίας κλπ. Ε, δεν μιλάμε για στρατιές ε, επιτόπου. Δεν θα υπάρξει αυτή η περίπτωση. Τώρα, ερχόμενοι. Τώρα στο, στο ερώτημα της κυρία Νικολά. Σύμφωνο βεβαίως ότι η διαφθορά είναι πρόβλημα σε μερικές από αυτές τις χώρες. Ε, και ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο ρόλος του στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας μειώνεται, αποδυναμώνεται από, τα, από τις προσόδους και τα ωφέλη των παρανόμων ε, ενεργειών. Είναι λοιπόν πράγματι ένα στοιχείο αυτό και γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ασφάλεια, διότι δεν μπορεί κανείς ε, να καταπολεμήσει τη διαφθορά εάν δεν μπορεί να εδρεώσει τα, ε, τους θεσμούς, παραδείγματος χάρη την απονομή της δικαιοσύνης, η λειτουργία του κράτους κλπ. Για τους πρώην φόρους τις, ε, τις στρατιώτες ή τις δυνάμεις στρατιωτικές στην Λιβύη, εμείς δεν ε, προσεγγίζουμε το όλο θέμα ως ε, τόσο απειλητικό. Οι περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις, οι μισθοφόροι προέρχονται από στρατιωτικές δυνάμεις είτε του Νίγηρα είτε του Μαλή και μπορεί να επιρέτησαν ως μισθοφόροι ένα χρονικό διάστημα αλλά εν συνεχεία γυρίζουν πίσω, επανέχουν στις δικές τους δυνάμεις. Ε, ε, ορισμένοι από αυτούς μπορεί ίσως να παραμείνουν ε, και να σηκώσουν και πάλι τα όπλα, ας πούμε, υπέρ του παλαιού καθεστώτος, αλλά... Πιστεύω ότι οι περισσότεροι, εάν τους δοθεί μια ευκαιρία, οι περισσότεροι δηλαδή από αυτούς τους πρώην μισθοφόρους που θέλουν να παραμείνουν, θα θέλουν να παίξουν ένα ρόλο, εάν τους δοθεί αυτή η ευκαιρία κυρίως από τον Ήγηρα προέρχονται και από το Μαλή Μερική, αλλά κυρίως στον Ήγηρα. Ακόμα και στον τομέα της ασφάλειας ενδέχεται ίσως στην αστυνομία, στην τοπική αστυνομία ή στο στρατό να μπορούν να ενσωματωθούν. Ε, κατά τα άλλα υπάρχει ένας κίνδυνος, αλλά υπάρχουν και άλλα, άλλες πτυχές τις οποίες πρέπει να εξετάσουμε για να αμβλύνουμε το τυχόν πρόβλημα. Ε, α, άλλες, άλλους τομείς ε, που συζητήσαμε σήμερα είναι η οικονομική ενίσχυση της ασφάλειας, αλλά όπως είπε και ο κύριος ε, Κερκόφ, δεν είναι τόσο πολύ θέμα χρημάτων έτσι καλώ τα χρήματα που έχουν δοθεί, τα 400 εκατομμύρια συν 150 εκατομμύρια ευρώ επαρκούν αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι είναι κατάλληλο το ποσό αυτών και οι χώρες του Μαγκρέπ ε, ήδη έχουν και αυτές λάβει πιστώσεις 150 εκατομμυρίων και πιστεύω ότι είναι πρόθυμες να συνεργαστούν στην ασφάλεια, στον τομέα της ασφάλειας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι παρεμβάσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση την οποία κάνατε, για την επικαιρότητα όλων αυτών των ζητημάτων. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την τακτική αυτή επαφή. Κάτι τελευταίο έχω να πω. Αναφερθήκαμε στις δραματικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών, ιδίως στο Μαλί. Μήπως έχετε περισσότερες πληροφορίες να μας δώσετε για τα γεγονότα αυτά. Όχι. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν σήμερα το απόγευμα στις 2.30 το μεσημέρι για την ακρόαση την οποία έχουμε όσον αφορά την, το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθε εντό των ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη και θα μιλήσουμε επίσης και για την Ευρωπαϊκή Διοίκηση Αερομεταφοράς. Ευχαριστώ πολύ.